Καλώς Καλώ ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι στη συνεδρία τη Επιτροπή Περιβάλλοντο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά κάποιοι γεωργοί με εμπόδισαν να έρθω και ήρθα λιγάκι αργότερα από ό,τι ήθελα να είμαι. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ που είσαστε εδώ στη συνεδρίασή μα. Πρώτο σημείο έγκριση τη ημέρησια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσει έχει εγκριθεί. Σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου, του υποφαινομένου. Έχω να σας πω κάτι σε σχέση με αυτά τα θέματα τώρα. Έχουμε μια ομάδα επισκεπτών από τη Βόρεια Ιλανδία, τους οποίους καλωσορίζω ένθερμα στην Επιτροπή μας. Και περνάμε στο πρώτο ουσιαστικό σημείο της σημερινής συνεδρίασης, την ε, ανταλλαγή απόψε με την Κατρίν Ζεσλέν Λανέλ, που είναι Γενική Διευθύντρια της ΕΑΤ, δηλαδή της Αρχής για την Τροφιμική Ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστή ως ΕΦΣΑ. Καλώς ήρθατε κυρία Λανέλ, Ζεσλέν Λανέλ, στην Επιτροπή μας, στο μόλις επανεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που με πολύ ενθουσιασμό και φυσικά με τον ενθουσιασμό των νέων μελών αλλά και των παλαιών θέλει να ανταλλάξει απόψη μαζί σας και υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν θέλω να χάσω όλο χρόνο, σας δίνω μέσα στο λόγο. Είμαι ευγνώμων για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας ενημερώσω για τις δραστηριότητες ε, της ε, υπηρεσίας Να σας συγχαρώ και για τις δραστηριότητές σας από εδώ και πέρα. Κυρίως να σημειώσω τις ευχές μου ε, και κάθε επιτυχία στη νέα σας εντολή. Αυτή στιγμή που ξεκινάει το νέο κοινοβούλιο συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και γενικότερα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Σαν υπεύθυνη υπηρεσία για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζω να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συλλογικές προκλήσεις. Η εμφάνισή μου σήμερα εδώ μου δίνει τη δυνατότητα να σας ενημερώσω για τα βήματα προόδου ε, τα οποία έχουμε κάνει. Είναι θα έλεγα και χρήσιμη γιατί μπορεί να θυμίσει ότι η υπηρεσία μου είναι στη διάθεσή σας και είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνετε με ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές. Επιμένω στις λέξεις επιστήμη και στη λέξη επιστημενικός στο επίθετο επιστημονικός, γιατί αυτή είναι η δουλειά την οποία κάνουμε και σε καμία περίπτωση εμείς δεν λαμβάνουμε αποφάσεις που ναύτονται της πολιτικής. Η υπηρεσία μας, η υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων, δημιουργήθηκε το 2002 με στόχο να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επιστημονική βάση για τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει στον συγκεκριμένο τομέα και διευκολύνουμε επίσης και την επικοινωνία στους κινδύνους που αφορούν στα τρόφιμα και την τροφιμική αλυσίδα. Ε, καθοδηγούμενοι από τον ιδρυτικό μας κανονισμό προσπαθούμε να λειτουργήσουμε επί τη βάση των κριτηρίων των, της επιστήμης, της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκομένους. Τη τελευταία δεκαετία ζήσαμε πολλούς φόβους στον τομέα των τροφίμων και αυτό απαιτεί να διαχειριστούμε τους κινδύνους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το τρόπος αυτός, το πρότυπο αυτό, έχει βοηθήσει έτσι ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των εμπορικών μας εταίρων στα τρόφιμα τα οποία διαθέτουμε. Η διαθεσιμότητα της εμπειρογνωμοσύνης αυτής ε, διαπερνά θα έλεγα πολλούς επιστημονικούς τομείς και έχει πολύ μεγάλη σημασία για την υπηρεσία μου έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ερωτήσεις τις οποίες μαθαίνουν αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τον κίνδυνο. Χρησιμοποιούμε την εμπειρογνωμοσύνη 1.500 επαϊόντων στο σύνολο της Ευρώπης, οι οποίοι προσφέρουν, θα έλεγα, τον χρόνο τους για την προστασία του Ευρωπαίου καταναλωτή. Μέσω της επιστημονική μας επιτροπής και των 10 επιστημονικών πάνελ, η υπηρεσία μας δίνει την δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες των διαχειριστών κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ασχολούμεθα με θέματα υγείας επίσης και κτηνιατρικού τύπου, και όλο και περισσότερο καλούμεθα να εργαστούμε σε τομείς οι οποίοι δεν θεωρούνται παραδοσιακά ανήκοντες στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Κάποιος από το κοινό που βλέπει τις ε, γνωμοδοτήσεις που παράγουμε, γιατί, ε, αναρωτιέται γιατί ασχολούμεθα με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή την αποτελεσματικότητα των, εντομο, των εντομοκτώνων. Παρ' όλα αυτά, ο τομέας της ασφάλειας τροφίμων είναι ευρύτατος η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον συνδέονται πάρα πολύ στενά και η αηφορία των πρακτικών παραγωγής τροφίμων έχει κεφαλαιόδη σημασία για όλους. Η συνεργασία με τα κράτη-μέλη είναι κεντρική επίσης και για τη δυνατότητα που έχουμε να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Και γι' αυτό ακριβώς συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη σε όλα τα επίπεδα. Η σημασία της συνεργασίας υπογραμμίζεται κυρίως κατά τη διάρκεια επιγουσών καταστάσεων. Σαν παράδειγμα, η επιθυμία των Ιρλανδικών αρχών να μοιραστούν μαζί μας δεδομένα και πληροφορίες είναι κάτι το οποίο μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το ατύχημα με τη διοξίνη το 2008. Οι δομές μας είναι πλέον καθορισμένες. Υπάρχει Συμβουλευτική Επιτροπή, το Συμβουλευτικό Φόρουμ περισσότερο, το οποίο συγκεντρώνει εκπροσώπους από τις 27 εθνικές ανεξάρτητες αρχές ασφάλειας τροφίμων. Βασική μας προτεραιότητα είναι η ανταλλαγή επιστημονικής πληροφόρησης και επικοινωνία στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου. Άνω των 300 ευρωπαϊκών οργανώσεων συνεργάζονται μαζί μας και το 2009 χρηματοδοτήσαμε προγράμματα στα διάφορα κράτη-μέλη σε ύψος 7 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της προσπάθειάς μας που στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής είναι να, οδηγήσουμε, να οδηγηθούμε μάλλον σε μια δυνατότητα ε, συνολικής και ολοκληρωμένης μορφής αντίληψης και διαχείρισης του κινδύνου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Οι, πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει να χρησιμοποιηθούν με πολύ προσεκτικό τρόπο. Προσπαθούμε επίσης να αποκαταστήσουμε λειτουργικές σχέσεις με τις αδελφές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον έλεγχο των πανδημιών και των ασθενειών. Ε, ασχολούμεθα με θέματα όπως η αντίσταση στα αντιμικροβιακά και στα αντιβιωτικά και ασχολούμεθα επίσης και με τις ζωονόσους. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών. Η υπηρεσία μας λοιπόν σήμερα είναι μια όρημη οργάνωση με 450 άτομα προσωπικό. Δύο τρίτα από αυτούς εμπλέκονται σε επιστημονικές δραστηριότητες. Προσπαθούμε ε, να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας μας και να είμαστε εξοπλισμένοι ώστε να δίδουμε έγκαιρα και με εύθετο τρόπο την επιστημονική μας συμβουλή. Προσπαθούμε να προλάβουμε τις αλλαγές στην νομοθεσία και γι' αυτό ο διάλογος με τις πολιτικές αρχές μαζί σας συγκεκριμένη περίπτωση είναι κρίσιμος. Η προσπάθεια την οποία κάνουμε σε σχέση με τις αιτήσει για αδειοδότηση είναι μια δραστηριότητα η οποία δεσμεύεται χρονικά θα έλεγα, καταναλώνει το 35% των πόρων μας. Αυτές οι αιτήσει για αδειοδότηση έχουν σχέση με τρόφιμα, με πρόσθετα τροφίμων, αρωματικές ουσίες, ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ε, υλικά ε, πακεταρίσματος, εντομοκτώνα, καινοτόμα τρόφιμα και ήδη την προηγούμενη εβδομάδα θα έλεγα δημοσιεύσαμε 94 γνωμοδοτήσεις για 523 αιτήσει πιθανής ανομαλίας στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας δώσει απαντήσεις για 2.000 περιπτώσεις, τις οποίες ζητήθηκαν επιπλέον πληροφορίες και έχουμε λάβει επίσης και 500 νέες αναφορές. Σε σχέση με αυτό τον όγκο δουλειά, θα έλεγα μόνο ότι δείχνει την μεγάλη σημασία που ο κόσμος θεωρεί ότι πρέπει να έχουν οι εργασίες μας. Έχουμε και το πάνελ μας σε σχέση με τα διαιτητικά προϊόντα και τις αλλεργίες. Έχει και άλλες ε, δραστηριότητες σημαντικές, βοηθώντας ε, αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο ε, να αποφασίζουν για θέματα όπως η υγιεινή τροφή, η μείωση επίσης των υπέρβαρων Ευρωπαίων πολιτών. Το 2010 θα δημοσιεύσουμε περισσότερο στοιχεία για τις λεγόμενες μακροτροφημικές ουσίες οι οποίες θα βοηθήσουν τους ε, διαχειριστές του κινδύνου να καθορίσουν κατευθυντήριες κατάλληλες γραμμές. Ήδη από το 2009 ο αριθμός ε, ε, των συνεργατών, των αναφορών τις οποίες δημοσιεύουμε θα αυξηθεί πολύ περισσότερο από τις 500 επιστημονικές αναφορές τις οποίες δημοσιεύσαμε το 2008 απαιτείται ποιότητα, απαιτείται εύθετος χρόνος ανταπόκρισης, αυτά είναι καθοριστικά για την αξιοπιστία της υπηρεσίας μας και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει και με το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας για την επιστημονική παραγωγή μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμεθα με επάρκεια και με ταχύτητα στα κατεπήγοντα θέματα. Μας έχει ζητηθεί να δράσουμε με μεγάλη ταχύτητα, δίδοντας σύμβουλες και συστάσεις έτσι ώστε να μην ζήσουμε κρίσεις όπως αυτές της δεκαετίας του 1990 που απειλούν τη δημόσια υγεία και διαρριγνύουν τις εμπορικές ροές. Θέματα όπως η μελαμίνη στα τρόφιμα είναι θέματα στα οποία αντιδράσαμε μέσα σε μέρες και όχι σε μήνες και ακριβώς αυτή η ταχύτητα βοήθησε και τους πολιτικούς να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. Οι συστάσεις τις οποίες δίδουμε στους νομοθέτες θα επηρεάζουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών και ακριβώ μέσω των πρωτοβουλειών διαβούλευση, τι οποίε αναλαμβάνουμε καλύπτουμε το σύνολο των εταίρων στην τροφιμική αλυσίδα. Ε, συμπεριλαμβάνουμε στις διαβουλέσεις αυτές ε, και ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος και ομάδες καταναλωτικές. Καλύπτουμε τομείς όπως οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, η κλωνοποίηση, πολύ σημαντικούς τομείς στους οποίους υπάρχουν και πολύ σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους εταίρους. Σε αυτή τη φάση ανανεώνουμε τα μέλη της ε, πλατφόρμας ε, της συμβουλευτικής που έχουμε για τους εμπλεκομένους φορείς, που περιλαμβάνει γεωργούς, ε, την βιομηχανία τροφίμων, την βιομηχανία διανομής, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών κτλ. Η υπηρεσία μας προσπαθεί να βελτιώσει την ικανότητά της να επικοινωνεί και έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου, αλλά αυτό δεν φτάνει. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας με ε, όλα τα επίπεδα με τα οποία ε, έχουμε μια κάποια ανταπόκριση. Το 2008 ήμουν εδώ παρούσα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος στα πλαίσια του στρατηγικού προγράμματός μας για την περίοδο 2009-2013 και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Το πρόγραμμα αυτό υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαίος σήμερα στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα και η τελική απόφαση ελήφθη από τη διαχειριστική μας επιτροπή το Δεκέμβριο του 2008 και είμαστε τώρα στη φάση εφαρμογής. Αυτή είναι και η βάση για τα ετήσια προγράμματα εργασίας μας και ε, το πρόγραμμά μας για το 2010 είναι ήδη γνωστό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει δύο βασικές πρωτοβουλίες για το 2010, οι οποίες είναι σημαντικές για την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιολογεί σωστά τους κινδύνους και για την προσπάθεια αυτή η δική σας στήριξη είναι απαραίτητη. Η πρώτη από τις δύο αυτές πρωτοβουλίες έχει σχέση με τη συλλογή των πληροφοριών και την ανάλυση τους. Η δυνατότητα συλλογή των δεδομένων είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει το σύνολο των εργασιών μα. Το 2009 δημοσιεύσαμε εννέα μείζονε εκθέσει για τα θέματα τη επιμόλυνση επιμόλυνσης των τροφίμων. Τον Μάιο δημοσιεύσαμε την Συνολική Επιτροπή to monitor salmonella reduction programs για ασθένειε, οι οποίε προκαλούνται από τα τρόφιμα, μέσω των τροφίμων και διαδίδονται μέσω των τροφίμων όπω η σαλμονέλα. Έχουμε δώσει στοιχεία τα οποία θα χρησιμεύσουν για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα σας στείλουμε επίσης και μία έκθεση για τη συλλογή δεδομένων για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών που θα περιγράφει την σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη εντοπίζοντας πιθανές αδυναμίες και κάνοντας συστάσεις για βελτιώσεις. Μπορώ να σας πω από τώρα ότι η έκθεση αυτή εντοπίζει την επίγουσα ανάγκη για μια πανευρωπαϊκή ε, προσπάθεια, μια ενιαία ευρωπαϊκή προσπάθεια, έτσι ώστε τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε να είναι πράγματι ιδιαίτερος αξιόπιστα. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε σωστά τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται ο καταναλωτής μας και ε, για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε τι τρώγει φυσικά αυτός ο καταναλωτής. Τα δεδομένα δεν είναι συγκρίσιμα και δεν προέρχονται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα κράτη-μέλη και δεν είναι όπως είπα ακριβώς συγκρίσιμα η πανευρωπαϊκή έκθεση αυτή για την κατανάλωση τροφίμων, την οποία σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε το 2010, θα μας δώσει επιπλέον στοιχεία και θα έχει και άλλες δυνατές εφαρμογές, όπως τον τομέα της διατροφής γενικότερα, όπου τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ε, σύσταση συγκεκριμένων μορφών διατροφής που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα μια τόσο μεγάλη προσπάθεια η οποία θα έχει τόσο απτά αποτελέσματα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή απαιτεί φυσικά πάρα πολύ σημαντικούς πόρους. Και ενώ από τη μία η υπηρεσία μας είναι διατεθειμένη και πανέτοιμη να χρησιμοποιήσει τους πόρους τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, θα απαιτηθούν περαιτέρω συνεισφορές και από τα κεντρικά ευρωπαϊκά ταμεία αλλά και από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενισχύσει την πρωτοβουλία αυτή και την εταιρική σχέση. Η δεύτερη κεντρική πρωτοβουλία μας για το 2010 συνδέεται με, την, με τον εντοπισμό και την ανείχνευση των ε, κινδύνων που βρίσκονται σε διαδικασία εμφάνισης των αναδυόμενων κινδύνων. Πρέπει η Ευρώπη να μπορεί να αντιδράσει ε, ταχύτατα σε τέτοιου είδους μορφές κινδύνου και να προσπαθήσει να λειτουργήσει προληπτικά. Γι' αυτό ακριβώς θα παρουσιάσουμε την πρώτη ετήσια έκθεση για τους αναδιόμενους κινδύνους στα τρόφιμα στην Ευρώπη στις αρχές του 2010. Η εμπιστοσύνη στην τροφιμική μας αλυσίδα είναι κάτι που πήρε πάρα πολλά χρόνια για να οικοδομηθεί, αλλά όπως έχει μάθει η Ευρώπη με οδυνηρό τρόπο μπορεί να καταστραφεί η εμπιστοσύνη αυτή με ένα συγκεκριμένο ατύχημα. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες μας στον τομέα της πρόβλεψης και πρόληψης, έτσι ώστε να μπορέσουμε νωρίς και σε έφετο χρόνο να ανταποκριθούμε ε, αντιμετωπίζοντας τις περιπλοκές που μπορεί να επιφέρει η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, οι κλιματολογικές αλλαγές και η τεχνολογική καινοτομία. Η συνεργασία αυτή απαιτείται να γίνεται σε παγκόσμιο φυσικά επίπεδο με τις επιστημονικές μας επιτροπές και τα επιστημονικά πάνελς, η υπηρεσία την οποία έχουμε για την αξιολόγηση των αναδειωμένων κινδύνων προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες πολλών περιοχών διαφορετικών μεταξύ τους στο σύνολο της Ευρώπης και πέραν αυτής. Συμπερασματικά, απαιτείται να συνεχιστεί η υποστήριξή σας ιδιαίτερα για τα δύο αυτά κομβικά προγράμματα για το 2010. Θα προσφέρουν ιδιαίτερα ωφέλη στον Ευρωπαίο καταναλωτή και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών μας. Είναι μεγάλη τιμή για μας να σας δείξουμε από κοντά τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας προσκαλέσω στα γραφεία μας στην Πάρμα της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση θα θέλατε να μου θέσετε. Ναι, ευχαριστώ κυρία Ζησλέν Ντανιέλη. Ε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Πραγματικά, από το 2002 έχει ανθίσει, έχει αναπτυχθεί ε, η προσπάθειά σας, το Κοινοβούλιο πάντα ανταποκρινόταν στις επιθυμίες σας και για το προσωπικό και τις οικονομικές και πάλι είπαμε βεβαίως ότι θέλουμε να συνεχίσει τη δουλειά σας. Έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι. Ο Ρίχαρτ Ζέμπα πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία Γενική Διευθύντρια, σας ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, η ασφάλεια τροφίμων και η σχέση με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς είναι ένα θέμα πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο και απασχολεί πάντα τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει δοθεί καμία άδεια ε, μάλλον δεν έχει ε, υποβληθεί καμία αίτηση για άδεια ε, προϊόντος ή για ουσίες που να έχει απορριφθεί. Όλες οι αιτήσει που υποβάλλονται εγκρίνονται. Παρ' όλα αυτά οι επιστήμονες δηλώνουν ότι είναι ενδεχομένως επικίνδυνες. Εσείς τι λέτε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε σύντομα πώς λαμβάνετε τις αποφάσεις και μέχρι τώρα γιατί δεν λαμβάνετε υπόψη και τις αρνητικές μελέτες, δεν βρίσκουν το δρόμο τους στις, προς τις αποφάσεις σας αυτές ή λίγο. Και μια ε, δεύτερη ερώτηση για τον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα Novel Food. Είναι ένα θέμα με το οποίο συνεργάζεστε, ε, με, με, μάλλον έχετε ένα προγραμματισμό να συνεργαστείτε με το ε, Αμερικανικό αδελφό οργανισμό Food and Drug Administration αλλά εμείς έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, όπως γνωρίζετε, ε, που πρέπει να σας μεταφέρουμε, ανησυχίες και επιφυλάξεις των πολιτών. Και μια τελευταία ερώτηση για τα νάνο υλικά. Τι έχουμε εκεί από εκτίμηση κινδύνου. Είναι μια ε, πολύ ελπιδοφόρα τεχνολογία και έχει βρει το δρόμο της ήδη προς τα ε, τρόφιμα. Μπορείτε να μας πείτε πώς έχουν εκεί τα πράγματα. Ευχαριστώ, Ελίντα Μακάβαν. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Διευθύντρια της ΕΦΣΑ για την παρουσία της στην συνεδρίασή μα. Προσβλέπω σε μια συνεργασία μαζί σας στο νέο Κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε την πρόοδο σε σχέση με τις αγωγέ που έχουν συγγνώμη, σε σχέση με τους ισχυρισμού για το υγιεινό των τροφίμων και νομίζω με τον τρόπο αυτό μπορούμε να, εξαντλήσουμε να εξαλείψουμε μερικέ από τις πιο παραπλανητικές τέτοιε μορφέ ισχυρισμού. Τώρα, στον τελευταίο κανονισμό που εγκρίναμε με το Συμβούλιο, θέλαμε να εξαλείψουμε τρόφιμα τα οποία έχουν υπερβολικό περιεχόμενο άλατος και συγχρόνως συνοδεύονται από ισχυρισμούς υγιεινότητας. Και θέλαμε να έχουμε ένα προφίλ για τα υγιεινά τρόφιμα, ώστε να αποφύγουμε τέτοιες περιπτώσεις. Θα ήθελα να ξέρω τι συμβαίνει σε σχέση με αυτό το θέμα, γιατί ανησυχώ λιγάκι. Τις τελευταίες εβδομάδες μου είπανε πολλοί ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν εκτροχιαστεί. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει πράγματα όπως το να επιτρέπει να θεωρούνται υγιεινές τροφές, να υπάρχουν ισχυρισμοί υγιεινότητες στροφών που δεν είναι καθόλου υγιεινές. Μέσα στις προτάσεις λοιπόν της Κομισιόν υπάρχουν τέτοιου είδους παραθυράκια. Ακόμα και τα παγωτά θα θεωρούνται υγιεινά. Το θέμα λοιπόν είναι δεν είναι αν θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να διατίθενται στο κοινό, αλλά αν θα πρέπει ορισμένοι να θεωρούν και να ισχυρίζονται ότι είναι υγιεινά. Δεν θέλω να ξέρω αν θα έχουμε κάποιε προτάσει λοιπόν από εσά σε σχέση με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο Chris Davis. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τονίσατε ότι ο στόχος της ΕΦΣΑ είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων, κατά κύριο λόγο. Το μεγαλύτερο μέρος όμως της εργασίας σας και η περιοχή ευθύνη σας έχει ξεπεράσει αυτόν τον τομέα. Ασχολείστε και με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Θα ήθελα εδώ να θέσω το εξής ερώτημα. Μέχρι πού φτάνετε. Παραδείγματο χάρη για το θέμα των μελισσών. Μπορείτε εσεί να θεωρηθείτε κριτής βιοπικιλότητα και μπορείτε να θεωρηθείτε ότι εσεί μπορείτε να στραφείτε εναντίον ορισμένων προϊόντων τα οποία δεν κάνουν κακό στον άνθρωπο αλλά μπορεί να κάνουν κακό στα έντομα όπως είναι Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι υπερβαίνετε την αρχική σας εντολή ως ΕΑΤ, ως ΕΦΣΑ, με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει τύχει επαρκούς ελέγχου μέχρι στιγμής. Λοιπόν, μέχρι πού φτάνουν τα όρια της αρμοδιότητάς σας σε σχέση με τέτοια θέματα, δηλαδή αν πρέπει να είσαστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της ποιότητας στην φύση εν γέννη και μήπως θεωρείτε ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα φορέων όπως ο Ευρωπαϊκός Φορέας για τις Χημικές Ουσίες ή ο Ευρωπαϊκός Φορέας για το Περιβάλλον. Καλύτερα. Ευχαριστώ. Η Σάντριν Μπελιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γεια σας κυρία Διευθύντρια. Θα ήθελα να επανέλθω στις τελευταίες αυτές εκτιμήσεις κινδύνου για ένα συγκεκριμένο είδος αραβόστου, του αραβοσίτου 810. Λέτε ότι οι οργανισμοί δεν είναι γενετικά τροποποιημένοι, μπορούν να έχουν κάποια προβλήματα, να δημιουργήσουν προβλήματα για την καλλιέργεια του αραβοσίτου. Αλλά στην Ευρώπη δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Τον Απρίλιο 2008 ζήτησε η Κομισιόν από την ΕΦΣΑ να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα σε άμεσο χρονικό διάστημα των μη κυβερνητικών οργανισμών και να διευρύνει τους, ε, τις γνώσεις της. Αλλά η ΕΦΣΑ δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει αυτή τη νομική υποχρέωσή της που είναι η εξέταση του αντικτύπου σε μακροπρόθεσμο επίπεδο μέσα στο περιβάλλον. Γι' αυτό θέτω τα εξή ερωτήματα. Πρώτον, συμφωνείτε ότι αυτή τη στιγμή οι μακροπρόθεσμες ε, συνέπειες της καλλιεργίας μη, κυβεν, μη ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών δεν μπορούν ακόμα να εκτιμηθούν και επίσης οι προσπάθειες για τον ε, αραβόσιτο Μονσάντο 810 δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα σε κάποιους οργανισμούς και μήπως θεωρείτε ότι αυτό είναι επαρκής λόγος για να μην εγκριθεί η καλλιέργεια του αραβοσίτου το 810. Ευχαριστώ. Τα είπατε πολύ γρήγορα και οι διερμηνείς ασθμένουν για να σας προλάβουν όταν διαβάζετε ένα κείμενο, τουλάχιστον να μην το μιλάτε με τόσο, να μην το αναφέρετε με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Ίσως μπορείτε να απαντήσετε, κυρία Διευθυντή. Σας ευχαριστώ. Σε σχέση σε σχέση με τις δραστηριότητες που έχουμε αναπτύξει στον τομέα των μη, μη των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών, πρέπει να σας πω ότι από τη δημιουργία της ΕΦΣΑ έχουμε αντιμετωπίσει 98 αιτήσει σε σχέση με μεταλλαγμένους οργανισμούς και έχουμε δώσει γνωμοδότηση για κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, επιστημονικές ε, γνωμοδοτήσεις. Από τις 98 αυτές τώρα περιπτώσεις που μας έχουν παραπεμφθεί, στην περίπτωση 8, 8 αιτήσεων, υπήρξε απόσυρση αυτών των αιτήσεων όταν εμείς ζητήσαμε περαιτέρω πληροφορίες. Έχετε δίκιο λοιπόν, όταν λέτε ότι εμείς δεν έχουμε δώσει ποτέ αρνητικές γνωμοδοτήσεις, αν αρνητική είναι μια γνωμοδότηση που λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον από μια καλλιέργεια. Αλλά είναι γεγονό ότι όταν ζητήσαμε πρόσθετε πληροφορίε από ορισμένου ετούντε, αυτοί προτίμησαν να αποσύρουν την αίτησή του. Κατά εμέ, αυτό σημαίνει ότι εμεί έχουμε ήδη εντοπίσει κάποια σημεία πιθανή ανησυχία και δεν θεωρούσαν ότι είχαν την δυνατότητα να συνεχίσουν τη διαδικασία Αξιολόγηση κινδύνου και μετά έγκριση για τα προϊόντα αυτά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό είναι το εξή. Σε, για 95% των αιτήσεων που λαμβάνουμε εμεί ζητούμε πάντα πρόσθετε πληροφορίε σε σχέση με την αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πραγματικά ενεργοί και εξασφαλίζουμε ότι μας δίδονται και πρόσθετες πληροφορίες για να έχουμε επαρκή έλεγχο αντικτύπου και αξιολόγηση κινδύνου. Αναφερθήκατε τώρα στη συνεργασία που έχουμε, όχι μονάχα για τα νέα τρόφιμα, αλλά γενικά με την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμακευτικών Ουσιών, την FDA. Μπορώ να διευρύνω ίσω το ερώτημά σας και να σας πω ότι θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα, διότι εμείς ω φορέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αναπτύξουμε συνεργασία με τους ομολόγους μας και σε άλλες υπήρους και σε άλλες χώρες για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης και επειδή θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να επηρεάσουμε και το έργο ομολόγων φορέων σε διεθνείς οργανισμούς. Και γι' αυτό εμείς συνεργαζόμαστε στα πλαίσια του Codex Alimentarius για να υποστηρίξουμε τη δράση της Κομισιόν, αλλά και στα πλαίσια του ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη κατευθυντηριών γραμμών για την αξιολόγηση των κινδύνων. Η Food and Drug Administration των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σημαντικό εταίρος για μας, όχι γιατί εμείς θα πρέπει να αντιγράψουμε την FDA να ευθυγραμμίσουμε το έργο μας μαζί τους, αλλά γιατί θεωρούμε ότι είναι πρόσφορο να συμμεριζόμαστε επιστημονικές πληροφορίες. Γι' αυτό το 2007 υπογράψαμε μια συμφωνία εμπιστευτικότητας με την FDA, και πιστεύω ότι έχουμε εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και έχουμε αποκομίσει θετικά αποτελέσματα στην περίπτωση τομέων όπως η νανοτεχνολογία ή η κλωνοποίηση, γιατί έχουμε πρόσβαση σε αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί μεν, είναι όμως διαθέσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, θεωρώ ότι είναι θετική συνεργασία μας με την ε, Food and Drug Administration και με άλλους φορείς για ένα ευρωπαϊκό φορέα, μια ευρωπαϊκή υπηρεσία όπως η ΕΦΣΑ είναι απαραίτητο να έχουμε πρόσβαση στα καλύτερα επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα και να έχουμε φυσικά και δυνατότητα να επηρεάσουμε το έργο άλλων φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο για τις νανοτεχνολογίες και τα νανοσωματίδια. Σίγουρα έχετε δίκιο όταν λέτε ότι αυτό είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας. Πήραμε πέρσι εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας να βοηθήσουμε για να εντοπίσουμε καλύτερα και ενδεχομένω να ε, χαρακτηρίσουμε τους ενδεχόμενους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να προκύψουν από τη χρήση της νανοτεχνολογίας στην, ε, στα τρόφιμα και την τροφική αλυσίδα. Έχουμε δώσει μια πρώτη γνωμοδότηση σε επιστημονικό επίπεδο. Είναι δύσκολος ο τομέας αυτός, γιατί είναι πολύ λίγα τα δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα για την πτυχή ασφαλείας και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον της χρήσης της νανοτεχνολογίας, Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το θέμα αυτό για να εξασφαλίσουμε το ότι θα είμαστε σε θέση να αρρωγήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την ε, ρυθμιστική διαδικασία στην οποία πρέπει να υπόκεινται οι νανοτεχνολογίε. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα όμω, Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχει πει η Επιστημονική Επιτροπή στην ΕΦΣΑ είναι ότι οι τοξικολογικέ μελέτε οι οποίε χρησιμοποιούνται κανονικά για άλλα πιο συμβατικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην περίπτωση προϊόντων που περιλαμβάνουν στοιχεία νανοτεχνολογίας αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε πιο συγκεκριμένη έρευνα και αξιολόγηση για όλα τα νανοσωματίδια. Έχουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Ένα αφορά στοιχεία υλικών για τη συσκευασία τροφίμων και εκεί αναφέραμε ότι για το συγκεκριμένο προϊόν ότι θα ήταν μάλλον απίθανο να προκύψει κάποιος κίνδυνος για τον καταναλωτή γιατί τα νανοσωματίδια δεν μπορούν να περάσουν από το υλικό συσκευασία στα τρόφιμα. Επίσης, υπήρξε μια άλλη αίτηση η οποία έχει να κάνει με τη χρήση νάνο σωματιδίων σε ζωοτροφές, όπου είπαμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αξιολόγηση κινδύνων. Για τους ισχυρισμούς υγιεινού χαρακτήρα των τροφίμων. Εσείς αναφερόσασταν κυρίως στο θέμα του προφίλ των θρεπτικών ουσιών. Εμείς έχουμε εκδώσει μια επιστημονική μελέτη, μια γνωμοδότηση μάλλον, και αυτή τώρα είναι η γνώση της Κομισιόν και των κρατών μελών, γιατί προφανώς δεν είναι η ΕΦΣΑ η οποία λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με το προφίλ των θρεπτικών ουσιών, εναπόκειται στα κράτη-μέλη, εναπόκειται και στην Κομισιόν να πάρουν τις αρμόδιες αποφάσεις. Εμείς αρρωγούμε την Κομισιόν για την προετοιμασία αυτού του προφίλ. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει στην ΕΦΣΑ για να ελέγξουμε και να δοκιμάσουμε το εφικτό διαφορετικών συστημάτων και μεθόδων για να αναπτύξουμε προφίλ θρεπτικών ουσιών. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω ευθέως το ερώτημά σας και δεν θα το απαντούσα το ερώτημα αυτό το αν κινούμεθα προς την σωστή ή στην λαθασμένη κατεύθυνση, αυτό πρέπει να το αποφασίσουν αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τους κινδύνους. Είναι γεγονός όμως ότι έχουμε δώσει τις επιστημονικές πληροφορίες στην Κομισιόν και εξακολουθούμε να τους βοηθούμε για την εξέταση του εφικτού του συστήματος αυτού. Αλλά οι διαχειριζόμενοι τον κίνδυνο είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν την τελική απόφαση για τα θέματα αυτά. <clears throat> Είναι επίσης ορθό το να πούμε ότι το έργο μας περιλαμβάνει όλο και περισσότερο περιοχές του επιστητού που δεν έχουν άμεση επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων, αλλά μπορεί να έχουν έμεση επίπτωση στα τρόφιμα. Γνωρίζετε ότι είναι αλληλοσυνδεδεμένο το περιβάλλον με την ανθρώπινη υγεία, ότι η ρήπανση του περιβάλλοντος μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων. Συγχρόνως, οι διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μέχρι στιγμής, εμείς έχουμε δράσει, όπως είπα και πριν, στο χώρο της ε, αξιολόγησης κινδύνων για το περιβάλλον, αλλά μέσα στα πλαίσια της εντολής μας. Εμείς δεν έχουμε φύγει, μέσα, έχουμε φύγει από τα πλαίσια της εντολής μας όπως αναφέρεται στον ιδρυτικό κανονισμό της ΕΑΤ. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς, όπου έχει ζητηθεί η ΕΦΣΑ, η ΕΑΤ, να, να παρέχει και αξιολογήσεις του αντικτύπου της καλλιεργίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον. Και ένα άλλο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι όταν εμείς εξετάζουμε αιτήσει για προσθετικά στα τρόφιμα, μας ζητείτε να αξιολογήσουμε και τον αντίκτυπο των προσθετικών αυτών για το περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, από πλευρά από πλευράς ρυθμιστικής δράσης μας, πρέπει να εξετάζουμε τον αντίκτυπο τοξικών ουσιών όπως είναι το κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα στην τροφιμική αλυσίδα. Και σε σχέση με τις μέλισσες που αναφέρατε, που μπορεί να είναι εκτός της εντολής μας, εδώ είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι, ότι η ζωή, η η υγεία των ζώων είναι μέσα στην εντολή της ΕΦΣΑ. Αυτό το είδαμε με τα προβλήματα με, την, με ασθένειες των ζώων στη δεκαετία του 1990. Ό,τι συμβαίνει στο αγρόκτημα, ό,τι συμβαίνει στα ζώα του αγροκτήματος και σε άλλα ζώα μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη δική μας ζωή, την ανθρώπινη ζωή και υγεία. Επομένως, είναι μέσα στην εντολή μας η υγεία των ζώων. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η χρήση παρασιτοκτόνων επίσης. Οι επιζωοτίες, κάποιες επιζωοτίες μπορεί να έχουν ε, επίπτωση στην υγεία των μελισσών. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει ένα σχέδιο συνεργασίας με ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτό ήταν αίτηση και της Κομισιόν και κάποιων κρατών μελών για να μπορέσουμε να, έχουμε, να έχουν αυτή μάλλον επιστημονική γνωμοδότηση και ανάλυση των δεδομένων τα οποία είχαν συλλέξει, κάτι το οποίο θα βοηθούσε τα κράτη-μέλη να εντοπίσουν καλύτερα τους λόγους για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, σημαντικά προβλήματα συγκεκριμένα, στον τομέα της μελισσοκομείας τα τελευταία χρόνια σε ορισμένα, αν όχι στα περισσότερα από τα κράτη-μέλη μας. Το γεγονός ότι έχουν καταρρεύσει οι απικίες μελισσών σε πάρα πολλές ε, χώρες, αυτό είναι μια ένδειξη του ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Γι' αυτό εργαζόμαστε και στον τομέα αυτό. για τον Μονσάντο 810, τον Αραβόστο. Εμείς ενημερώνουμε τακτικά τα έγγραφα κατεύθυνσή μας, όπως λέγονται. Είναι έγγραφα στα οποία εμείς και η επιστημονική ομάδα για τους μεταλλαγμένους οργανισμούς περιγράφουμε τη μεθοδολογία μας για την εκτίμηση του κινδύνου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να είναι γνωστό και να υπάρχει η πιο επακριβή συνατή περιγραφή του μηχανισμού και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούμε και για λόγους διαφάνειας, αλλά και για να μπορέσουμε να είμαστε ενήμεροι με τις τελευταίες επιστημονικές πρόοδους. Κάνουμε λοιπόν αυτή την τακτική ενημέρωση αυτών των εγγράφων μεθοδολογίας για την εκτίμηση κινδύνου και πέρσι συγκεκριμένα κάναμε μια αναθεώρηση σε σχέση με την εκτίμηση κινδύνων για το περιβάλλον που είναι τμήμα της συνολικής εκτίμησης κινδύνου που κάνουμε για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Και μας ζητήθηκε συγκεκριμένα να εξετάσουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών και να δούμε πώς μπορούμε <clears throat> να ενισχύσουμε την εκτίμηση κινδύνου στο μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ήδη λοιπόν περιλαμβάνουμε αυτό το στοιχείο στις αξιολογήσεις μας αλλά πρέπει να τονίσω ότι αυτό είναι και ένα πάρα πολύ δύσκολο τομέα. Όταν μιλάμε για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, σημαίνει αυτό ότι πρέπει να συλλέξει κανείς δεδομένα για την παρουσία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ένα μακρό χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χρονικό διάστημα εμπειρίας ίσως 10 χρόνων σε ό,τι αφορά την χρήση μεταλλαγμένων οργανισμών και όπως ξέρετε οι ετούντες και τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν και να αναπτύξουν προγράμματα εποπτείας του περιβάλλοντος για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Βάσει αυτών λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας για κάθε αίτηση εμείς μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση του αντικτύπου των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον αλλά περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να βελτιώσουμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε. Αυτό βέβαια είναι μια συνεχή διαδικασία. Αυτά που λένε σήμερα οι επιστήμονε, αύριο μπορεί να αποδειχθούν ότι είναι λανθασμένα. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε, να τροχοπεδίσουμε τη διαδικασία αξιολογήσεων, γιατί η επιστήμη είναι σε συνεχή αλλαγή και βελτίωση. Το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι βάσει αυτών τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας και μπορούμε απλώς να επισημάνουμε τις αβεβαιότητες που συνάπτονται με τις γνώσεις που έχουμε για να σας απαντήσω λοιπόν. Η ενημέρωση του εγγράφου κατευθύνσεων θα έχει σαν στόχο μεταξύ άλλων και το να ενισχύσουμε την ε, ε, εκτίμηση των επιπτώσεων των γενικά μεταλλαγμένων οργανισμών σε άλλους οργανισμούς εκτός, εκτός από αυτούς που είναι οι οργανισμοί στόχου, αυτοί οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα. Εν κατακλείδη λοιπόν, συνοψίζοντας, προφανώς θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο μας σε όλους τους τομείς και ιδίως σε αυτούς τους νέους τομείς όπως είναι η ανατοχνολογία, κλωνοποίηση, γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί, να βελτιώσουμε λοιπόν τη μεθοδολογία μας για την εκτίμηση κινδύνου αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους διαχειριστές κινδύνου και να γνωρίσουμε τι μπορεί να μας πει σήμερα η επιστήμη επί τη βάση των πληροφοριών που έχουν ήδη συλλέξει και αναλύσει. Okay. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις συνάδελφοι ακόμα. Η κάρτη Καλλιωτάς. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Κατρίν και σένα για τη παρουσία σου και την παρουσίασή σου. Καταρχάς, σε ευχαριστώ γιατί τα τελευταία δύο-δυόμιση ε, χρόνια που ήμουν εκπρόσωπος και σύνδεσμος ε, με την ΕΦΣΑ ε, λειτουργήσε πολύ καλά η συνεργασία. Θέλω να πω και στα νέα μέλη, αν έχετε απορίες και ερωτήσεις για την ΕΦΣΑ να απευθυνθείτε σε μένα. Γνωρίζω κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε πάντα, αλλά η επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αρκετά καλή. Ε, γνωρίζετε ότι συχνά είμαι και επικριτική. Θα σας κάνω και τώρα μερικές ερωτήσεις, αν δεν σας στεναχωρέσω και ελπίζω να μου απαντήσετε κιόλας. Ακούω ότι το τελευταίο καιρό ε, κυκλοφορούν διάφορες φήμες για μια πρόσθετη ουσία μόνο νάτριο γλουταμάτι, NSG, 621 βελτιωτικό της γεύσης είναι. Δεν ξέρω αν έχετε άμεση απάντηση να μου δώσετε. Αλλά θα ήθελα αν υπάρχει τίποτα να ενημερώσετε. Επίσης, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ορισμένα προβλήματα υγείας και αλλεργιών και κάποιοι κίνδυνοι. Εγώ δεν με, έχουν κάνει έρευνες δικοί σας της ΕΦΣΑ, αλλά υπάρχουν νέα στοιχεία, γίνονται νέες έρευνες και νέα δεδομένα. Έχω και άλλη ερώτηση για την κατάσταση του προσωπικού στην ΕΦΣΑ. Στην προηγούμενη θητεία ακούσαμε πολλές επικρίσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολλές ερωτήσεις. Βέβαια πάντα και οφείλω να το πω αυτό, ήταν πολύ καλή επικοινωνία και απάντηση της ΕΦΣΑ, αλλά στην τελευταία αλληλογραφία ρωτούσαμε αν μπορούσαμε να κάνουμε μια ανεξάρτητη έρευνα μεταξύ των μελών του προσωπικού για να δούμε πώς έχει η κατάστασή τους. Και μας απαντήσατε ότι ναι, αλλά το 2008 κάναμε μια τέτοια έρευνα που ε, έδειξε ε, ότι ανταποκρίνεται στα στάνταρ και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ειδικό λόγο να ρωτάει και ειδικό ερωτηματολόγιο για μια ειδική κατάσταση που έχει προκύψει. Και σας ερωτώ, θα γίνουν εξάρτητες τέτοιες έρευνες ε, στο προσωπικό σας μπορείτε να μας πείτε τίποτα παραπάνω τώρα για την κατάσταση ε, με τα διάφορα διατροφικά προφίλ. Και επίσης μας είπατε ότι θέλετε να κάνετε μια έρευνα για την ασπαρτάμι. Έχει προκύψει τίποτα καινούριο εκεί. Ε, και θα ε, περίμενα έτσι με μεγάλη ανυπομονησία και ενδιαφέρον να μας πείτε για την ασπαρτάμι. Ευχαριστώ. Ναι, ήσασταν ο σύνδεσμό μας με την ΕΦΣΑ και σα ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνετε τα τελευταία χρόνια. Πολύ χρήσιμη. Η κυρία Γκρουστέτ είναι η επόμενη συνάδελφος που έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μεγάλη χαρά, κυρία Διευθύντρια, να σας ξαναβλέπουμε στην Επιτροπή μας. δώσατε ήδη κάποιες απαντήσεις σε θέματα τα οποία μας αφορούν όλους. Θα ήθελα να επανέλθω στον κανονισμό σχετικά με τα καινοτόμα τρόφιμα. Στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης αυτών των φαρμάκων, εσείς παίζετε τον κεντρικό ρόλο. Εσείς ασκείτε, θα έλεγα, την δυνατότητα αξιολόγησης. Ξέρουν ότι κάποια αιτήματα, είναι πολλά τα αιτήματα που δέχεστε κάθε χρόνο, είτε για φυσικά τρόφιμα τα οποία είναι ασυνήθιστα στην Ευρώπη αλλά που έρχονται από άλλες υπήρους, είτε πρόκειται για νέα τρόφιμα τα οποία παράγει η βιομηχανία τροφίμων και θα ήθελα να μάθω τι γίνεται με τη λεγόμενη επιταχυμένη διαδικασία για την κυκλοφορία αυτών των νέων τροφίμων. Αυτή η επιταχυμένη διαδικασία μπορεί να είναι σε δύο περιπτώσεις απαραίτητη. Πρώτον γιατί πράγματι είναι χρήσιμο να πει κανεί ότι η Ευρώπη δεν δίνει τη δυνατότητα κυκλοφορία σε ένα νέο τρόφιμο, είτε γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε την καινοτομία και δεν πρέπει να ε, τροχοπεδούμε την ε, καινοτομία. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο για σας, είναι ένα επιπλέον, επιπλέον συγγνώμη βάρος στην προσπάθεια την οποία κάνετε. Έχετε συνεπώς τις δυνατότητες, έχετε τους πόρους που απαιτούνται για να καλύψετε αυτούς τους τομείς ευθύνης, για να αποφύγουμε τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Και πώς μπορείτε ε, επίσης να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία που έχουν οι εθνικές αρχές. Πώς ε, πηγαίνουν οι σχέσεις ανάμεσα στις εθνικές αρχές και εσάς στην Ιδία. Εσάς και την υπηρεσία σας εννοώ. Ευχαριστώ, κύριε Λεπάς. Ευχαριστώ την Διευθύντρια που είναι παρούσα σήμερα. Μία μικρή ερώτηση για τις νανοτεχνολογίες και με μια πιο σημαντική ερώτηση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Για τις νανοτεχνολογίες είπατε ότι έχετε αξιολογήσει δύο τέτοιες διαδικασίες. Μήπως είναι ανησυχητικό γνωρίζοντας ότι σήμερα υπάρχουν 150 τέτοιου είδους μόρια τα οποία χρησιμοποιούνται και στα τρόφιμα και στα καλλιντικά χωρίς να υπάρχει καν κατάλογος για να επιτρέψει στον Ευρωπαίο καταναλωτή να γνωρίζει τι καταναλώνει. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δύο σημεία. Το πρώτο αφορά τη μεθοδολογία και το δεύτερο την ουσία. Σχετικά με τη μεθοδολογία. Το Συμβούλιο Υπουργών, Υπουργών Περιβάλλοντος το Δεκέμβριο του 2008 αναφέρθηκε στις πρακτικές της υπηρεσίας σας σχετικά με την χρήση των επιστημονικών δεδομένων. Ε, τι ακριβώς συμβαίνει. Εσείς πιστεύετε ότι θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη μεθοδολογία τη συνενετική που δίνει συνεχώς ε, θετικές ε, γνωμοδοτήσεις. Τι γίνεται με τις μειονοτικές γνώμες. Μήπως θα πρέπει να κυκλοφορούν και αυτές έτσι ώστε να επιτρέπεται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να είναι σωστά ενημερωμένα. Για το 163 ε, είχατε εξετάσει για πρώτη φορά ε, το συγκεκριμένο αυτό γενετικά το αποποιημένο ε, φυτό. Μήπως θα πρέπει να βρείτε ένα διαφορετικό πάνελ και να δώσετε μια δεύτερη γνώμη. Τρίτον, σχετικά με τις ίδιες τις μελέτες τις οποίες προφαίνεται. Αν κατάλαβα αυτά που είπατε, οι μελέτες αυτές γίνονται ουσιαστικά από αυτούς οι οποίοι ζητούν τις αδειοδοτήσεις για γενετικά τροποποιημένους μηχανισμούς, οργανισμούς. Συγγνώμη. Μήπως θα ήταν προτιμότερο ε, να χρησιμοποιείτε ανεξάρτητους ε, επιστήμονες στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης γενετικά τροποποιημένων ουσιών και γενετικού υλικού κάτι το οποίο θα επιτρέψει στους επιστήμονες να λειτουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο, γιατί σήμερα, μιας και απαγορεύεται πλήρως για έναν ερευνητή το να έχει την δυνατότητα να αγοράσει σπόρους που θα του επιτρέψουν να κάνει ανεξάρτητες μελέτες, γιατί φυσικά οι σπόροι και η πώλησή τους ελέγχονται από τις εταιρείες και δεν θέλουν να χρησιμοποιηθούν. Μήπως οι σπόροι αυτοί Μήπως θα πρέπει να διευκολύνετε εσείς τις επιστημονικές μελέτες δίδοντας την πρόσβαση στη σπορία αυτή στους επιστήμονες. Σχετικά με τη μεθοδολογική πλευρά της εργασίας της. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο, ο εκμακρόθεν έλεγχος ξέρετε ότι δεν χρησιμοποιείται η χρήση των δορυφόρων κτλ. Η, ε, ο τηλεέλεγχος είναι κάτι το οποίο παραμένει μέχρι τώρα θα έλεγα στα ντουλάπια. Δεν είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως. Επιτρέψατε πρόσφατα τρία, τρεις νέους οργανισμούς γενετικά τροποποιημένους τρίτης γενεάς. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούν σπόρους ανθεκτικούς σε ε, εντομοκτώνα και γενικότερα σε ζυζανιοκτώνα. Ιδιαίτερα το 3022 ε, δεν έγινε αντικείμενο μελέτης επιποντικών σε, επιποντικών σε καμία περίπτωση. Πώς δίνετε εσείς ε, τέτοιου είδους άδειες κυκλοφορίες που χρησιμοποιούν ακριβώς ή μάλλον που είναι ανθεκτικοί σε ζυζανιοκτώνα και σε εντομοκτώνα χωρίς να ελέγξετε ε, την, ε, το παρελθόν τους σε πάση περιπτώσει. Είναι κάτι στο οποίο περιμένω την απάντησή σας. Γιατί το θέμα των εντομοκτώνων είναι κάτι το οποίο ε, συζητιέται όλο και περισσότερο. Και διαρωτώ με γιατί κάποιοι γενετικά τροποποιημένοι μηχανισμοί ανθεκτικής σε τέτοιου είδους ουσίες δεν δημιουργούν πρόβλημα, ενώ οι ουσίες οι ίδιες δημιουργούν πρόβλημα. Ιαν Ροσπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ε, πληρότητα των απαντήσεών σας και τα ενδιαφέροντα σχόλια σας, κυρία Διευθυντά. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα και τα ερωτήματα τα οποία σας ετέθηκαν. Θέλω λοιπόν να θέσω ένα ερώτημα το οποίο είναι κάπως κλασικού χαρακτήρα. Έχει να κάνει με την παραγωγή ζωοτροφών. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια προσθετική ουσία για τις ζωοτροφές και είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω έχει απασχολήσει το φορέα σας. Δεν ξέρω ποια είναι τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής της προσθετικής ουσίας στην υγεία των ζώων και στην ποιότητα του κρέατος και επίσης για τους καταναλωτές ποια είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μάθω σχετικά με το θέμα της ετικετοθεσίας που καλύπτουν τα λεγόμενα ασφαλή τρόφιμα. Δεν δίδουν οι ετικέτες αυτές όμως πληροφορίες παρά μόνο ιδιαίτερα ατελείς για τη σωστή διατροφή. Πώς μπορούμε εμείς να μην γίνεται μη υγιεινή χρήση υγιεινών κατά τα άλλα τροφών και πώς μπορούμε να ευνοήσουμε μια σωστή δίαιτα στον καταναλωτή γύρω από τρόφιμα τα οποία δεν είναι, δεν την χάνουν ετικετοθεσίας, φρούτα, λαχανικά, τα οποία δεν συνοδεύονται από ετικέτα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνει η δική σας υπηρεσία, αλλά νομίζω ότι είστε ο καλύτερος υποψήφιος για να προσπαθήσουμε να δώσουμε στον Ευρωπαίο πολίτη όλες τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να έχει στη διάθεσή του για μια ισορροπημένη δίαιτα. Και αναφέρομαι εδώ στην παχυσαρκία, ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κυρία Για, το μονονάτριο, για τη μονονάτριο γλουταμίνη, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς ξεκινάμε τη διαδικασία επισκόπησης της ε, ασφάλειας όλων των προσθετικών για τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια ε, έρευνα που έχει ζητήθει από την Κομισιόν και ξεκινάμε με τις χρωστικές ουσίες στα τρόφιμα. Και είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε την πρώτη μας γνωμοδότηση για τις πρώτες χρωστικές ουσίες τις οποίες έχουμε εξετάσει. Ίσως σας ενδιαφέρει ότι είναι έξι από τις χρωστικές ουσίες που αναφέρθηκαν στη μελέτη του Πανεπιστημίου του Southampton που δείχνουν κάποια δυνατότητα να υπάρχει κάποιο αντι... κάποιος αντίκτυπος. Η γλουταμίνη λοιπόν θα πρέπει να είναι μέσα στην αξιολόγηση αυτή των προσθετικών ουσιών και όταν γυρίσω στην Πάρμα θα, σας δώσω, θα μπορώ να σας δώσω πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για την προσθετική αυτή ουσία και κατά πόσο θα προκύψει μια επανεξέταση για το, την ουσία αυτή. Για το θέμα του προσωπικού της ΕΑΤ, της ΕΦΣΑ, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας ταχείας ανάπτυξης του φορέα μας. Είμαστε 450 μέλη του προσωπικού. Έχουμε φτάσει λοιπόν σχεδόν το μέγιστο επίπεδο οργανογράμματος που προβλέπετε. Πρέπει να προσλάβουμε ακόμα 20-30 μέλη του προσωπικού. Και έχουμε, πιστεύω προσέξει από την αρχή, για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε άτομα με υψηλά προσόντα σε επιστημονικό επίπεδο και επίσης και ικανότητα επικοινωνίας επειδή αυτό είναι πολύ σημαντικό για το έργο μας και το 2007 και 2008 ξεκινήσαμε να καταμετρούμε την ελκυστικότητα του φορέα μας τόσο για τα μέλη του προσωπικού γενικά όσο και ιδιαίτερα για τους εμπειρογνώμονες. Όπως και άλλοι φορείς, λοιπόν, κάθε χρόνο κάνουμε μια έρευνα μεταξύ των μελών του προσωπικού, κάνουμε και μια έρευνα των εμπειρογνωμόνων, γιατί όπως ξέρετε λειτουργούμε με ένα δίκτυο που περιλαμβάνει περίπου 1.500 εμπειρογνώμονες. Κάναμε λοιπόν αυτή τη μελέτη το 2008, τη δεύτερη έρευνα με ένα ερωτηματολόγιο περίπου 100 ερωτήσεων και θα επαναλάβουμε αυτό το εγχείρημα το Νοέμβριο εφέτος και το κάνουμε κάθε χρόνο για να μπορούμε να γνωρίζουμε αν εξακολουθούμε να είμαστε ελκυστικοί ως φορέας για την απασχόληση και τους εμπειρογνώμονες. Νομίζω τα πρώτα στοιχεία της προηγούμενης έρευνας ήταν θετικά. Αυτή είναι η εμπειρία μου λοιπόν ως ε, ε, διευθύντριες αυτού του οργανισμού. Περίπου 80% των μελών του προσωπικού μας ανέφερα μέσα στα πλαίσια αυτής της έρευνας ότι ήταν ευχαριστημένοι και ήταν υπερήφανοι να δουλεύουν για την ΕΦΣΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι εύκολα. Σίγουρα έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας στον οργανισμό μας. Ήταν στο παρελθόν ένας νέος οργανισμός και φυσικά πρέπει κανείς σιγά σιγά να δημιουργήσει μια κοινή κουλτούρα, μια κοινή αντιμετώπιση και επίσης θα έπρεπε να αναπτύξουμε μια πολιτική για τους ανθρώπινους πόρους και έχουμε πετύχει μια μεγάλη πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή και επίσης νομίζω ότι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής τουλάχιστον να διατηρήσουμε ένα λογικό ρυθμό ε, αντικατάσταση μέλλον του προσωπικού, δηλαδή να έρχονται και να φεύγουν ένα μικρό ποσοστό μονάχα. Και είμαι σε θέση να σας δώσω και άλλες ε, πληροφορίες, εάν θέλετε, μετά από την επόμενη έρευνα που θα ξεκινήσουμε σε λίγες εβδομάδες για την Ασπαρτάμι. Το 2008 είχαμε, είχαμε επιβεβαιώσει την ασφάλεια αυτού του, αυτής της γλυκαντικής ουσίας. Όπως γνωρίζετε όμως, αυτό ήταν ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέμα. Αυτή η προσθετική ουσία έδωσε λαβή σε πολλές διαμάχες και αποφασίσαμε, ιδίως ετήσι του Ηνωμένου Βασιλείου, να εξετάσουμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης και τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται ακόμα σε ορισμένα κράτη-μέλη δυνητικής ε, δυσανεξίας για την ασπαρτάμι ή άλλων μορφών αντικτύπου της ασπαρτάμις. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε λοιπόν να μας δώσει σε μας και στο δίκτυο των 27 εθνικών ομάδων εμπειρογνωμόνων τα στοιχεία αυτά. Το Νοέμβριο του ενεστώτος έτους θα συναντηθούμε και θα εξετάσουμε το θέμα αυτό και θα προκύψει και μια έκθεση η οποία θα είναι μια επιστημονική έρευνα η οποία θα είναι διαθέσιμη και στο ευρύ κοινό ώστε να μπορούν να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων αυτής της εξέτασης. Πιστεύω λοιπόν θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, όχι ότι έχουμε σημαντικές αμφιβολίες, αλλά σαν ένα ανοιχτό και διάφανο φορέας θεωρούμε ότι για ένα θέμα αμφιλεγόμενο όπω αυτό τη Ασπαρτάμη, να καταδείξουμε ότι εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τις περιπτώσεις οι οποίες ανέκυψαν σε ορισμένα κράτη-μέλη και να είμαστε ευαίσθητοι στις ανησυχίες του κοινού. Κυρία Γκροστέτ, ναι, για τα νέα τρόφιμα, ο κανονισμός αυτός φυσικά δημιουργεί πρόσθετο φόρτο εργασίας για την ΕΦΣΑ γιατί είναι πιο κεντρική η διαδικασία, συγκεντρωτική διαδικασία και έχουμε πιο στενά χρονοδιαγράμματα και επίσης γιατί η διαδικασία για τα νέα τρόφιμα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες οδηγεί και σε ένα νέο στοιχείο. Ότι δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να αντιστρέψουμε το βάρος της απόδειξης. Θα πρέπει εμείς να καταδείξουμε ότι υπάρχει ενδεχομένως αρνητικός αντίκτυπος στην υγεία, ενώ σε άλλους τομείς είναι ο ετών ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν είναι ασφαλές. Αλλάζει λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις αξιολογήσεις μας και έχουμε επομένως ένα πρόσθετο φόρτο εργασία για την ΕΦΣΑ. Εν γέννη και ιδίω για τα νέα τρόφιμα, νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι μας έχει υποστηρίξει η αρχή του προϋπολογισμού και ιδίω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω σκέλος αρχή αυτή του προπολογισμού. Νομίζω μέχρι στιγμή έχουμε τύχει τη πρέπουσα χρηματοδότηση. Αλλά θα έπρεπε να πω ότι όταν βλέπω την αύξηση του φόρτου εργασία μα, ιδίω σε ό,τι αφορά τα νέα νομοθετήματα τα οποία έχουν εγκριθεί, όπω πραγματικά χάρη αναφερθήκατε στα νέα τρόφιμα, αλλά πρέπει επίση θα, πρέπει να πούμε και για τα ένζημα, όπου περιμένουμε να υπάρξουν εκατοντάδε αιτήσεων προ την ΕΦΣΑ, τα FEE e και ενεργά υλικά συσκευασίας και εκεί περιμένουμε να λάβουμε αιτήσει σε σχέση με διαδικασίες ανακύκλωσης πλαστικών ουσιών, με τις προσθετικές επίσης ουσίες για τις, για όπου στα επόμενα τρία με 5 χρόνια θα πρέπει να επανεξετάσουμε 2.500 τέτοιες προσθετικές ουσίες. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Επομένως, νομίζω ότι είναι απαραίτητη η υποστήριξη της ΕΦΣΑ σε επίπεδο κονδυλίων. Εμείς προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των πόρων μας. Δεν ζητούμε μονάχα πρόσθετους πόρους, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μεγάλη πρόοδο στην εξέταση των αιτήσεων ώστε να είμαστε πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί όλο και περισσότερο εργαζόμαστε και με εθνικούς επιστημονικούς φορείς, όπως αναφέρατε. Συγκεκριμένα ζητούμε από εθνικούς φορείς ασφάλειας τροφίμων ή επιστημονικούς φορείς στα κρατη να μας αρρωγήσουν στο προπαρασκευαστικό μας έργο, ιδίως όταν πρόκειται για συγκεκριμένες αιτήσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία για μας είναι διαδικασίες που χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΦΣΑ. Αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι εάν συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλο και περισσότερες αιτήσει, στο μέλλον θα χρειαστούμε πρόσθετους πόρους. Εάν θέλουμε επίσης να εμπλέξουμε και περισσότερα κράτη-μέλη στο έργο μας, για να αναπτύξουμε την εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών αυτών, ίσως και εκεί πάλι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερα κονδύλια <clears throat> για την υποστήριξη των εθνικών φορέων και των εθνικών επιστημονικών οργανισμών νανοτεχνολογία και νανοσωματίδια. Έχουμε ήδη κάνει πολλή εργασία για τα θέματα αυτά. Έχουμε εξετάσει μονάχα νανοσωματίδια, τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ή σε διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών. Σε άλλους τομείς, και αναφερθήκατε ιδιαίτερα τα καλλιντικά, όπου υπάρχουν νανοσωματήρια στην αγορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας απασχολεί, δεν βρίσκεται μέσα στη δική μας αρμοδιότητα. Φυσικά, ίσως να μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τους τομείς αυτούς, όπως τα καλλινικά, γιατί και αυτό είναι χρήσιμο για την γενικότερη αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Εμείς όμως εξετάζουμε τα θέματα των σωματιδίων μονάχα στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και τις διαδικασίες παραγωγής των ανωτέρων. Για τους μεταλλαγμένους οργανισμούς έχετε αναφέρει πολλά σημεία. Εγώ ξεκινώ με την ε, σύσταση του Συμβουλίου το 2008, <clears throat> όπου το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, διατυπώνει την σύσταση για την αξιολόγηση κινδύνου που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριμένα για το έργο του δικού μας φορέα. Εξετάσαμε προσεκτικά αυτή την σύσταση του Συμβουλίου και η δική μας ανάγνωση είναι καταρχήν ότι υποστηρίζει το έργο της ΕΦΣΑ, δεν λέει ότι όλα είναι τέλεια, αλλά σίγουρα υποστηρίζει το έργο μας και ιδίω υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου της επιστημονικής αξιολόγησης κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον στον τομέα αυτό. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας. Αλλά επίσης αντιμετωπίζουμε και ορισμένες συστάσεις του Συμβουλίου, ιδίως δύο τέτοιες σημαντικές συστάσεις για το έργο μας. Μας ζήτησαν να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια της εργασίας μας. Κάνουμε όλο και περισσότερες προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Και σαν παράδειγμα μπορώ να σας πω ότι στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου εφέτος διοργανώσαμε εδώ στις Βρυξέλλες μια διάσκεψη με επιστήμονες από διάφορες προελεύσεις, είτε μέλη των επιστημονικών μας πάνελ, αλλά επίσης και εμπειρογνώμονες από κράτη-μέλη, οι οποίοι εμπλέκονται σε διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου για μεταλλαγμένους οργανισμούς, εμπειρογνώμονες από, το, από τη βιομηχανία και από μη κυβερνητικού φορείς όπως η Greenpeace, η φίλη της γης, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος κτλ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συνάντηση που κάναμε στην Πάρμα την ε, Παρασκευή με την παρουσία της Greenpeace και των φίλων της γης για να συζητήσουν μαζί μας και με τα μέλη του πάνελ για, την, ε, για τον Μονσάντο 810 που είναι ε, ένα προϊόν για το οποίο έχει γίνει αίτηση στην ΕΦΣΑ αξιολόγησης και μπορέσαμε να συζητήσουμε τα σχόλια αυτών των οργανισμών μαζί μας Επίσης τον συστήσαμε για τον οργανισμό NERAIS 62, για τον οποίο υπήρξε κάποια σύγχυση, κάποια σάφια σε σχέση με τη σύσταση που κάναμε για την ανάγκη ενός προγράμματος εποπτείας και παρακολούθησης αυτού του φορέα. Και εδώ είναι σαφές ότι πρέπει να καταβάλουμε όλο και περισσότερες προσπάθειες και φυσικά να καταβάλει προσπάθειες και ο διαχειριστής κινδύνου γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη συλλογή δεδομένων στα πλαίσια της διαδικασίας παρακολούθησης. Επίσης, συζητήσαμε με τους φίλους της γης και την Greenpeace τον τρόπο λειτουργίας μας και τις συστάσεις που έχει κάνει το Συμβουλίο σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων. Μία ακόμα σημαντική σύσταση που διατυπώθηκε από το Συμβούλιο αφορά τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη. Θα γνωρίζετε ίσως <clears throat> ότι για τον ΜΟΝ 810, τον Αναβόστο, είχαμε διάφορες ρήτες διαφύλαξης. Εμείς εξασφαλίσαμε ότι έχουμε ένα σωστό διάλογο με τους εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη και λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι οι επιστημονικές μας γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να εξετάζουν και να αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα σημεία τα οποία έφτιαξαν οι εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μας έχουμε τώρα σε ένα μακροσκελές παράρτημα, το παράρτημα G, την συμπίληση όλων των σχολείων που έχουν προκύψει από του εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, στα οποία σχόλια εμείς απαντούμε ένα προς ένα. Στο έργο μας επίσης, και πάλι αυτό αφορά τους μεταλλαγμένους οργανισμούς, αλλά επίσης και τους άλλους τομείς στους οποίους εμείς είμαστε ενεργείως φορέας, εμείς προσπαθούμε πάντα να περιλαμβάνουμε και τις απόψεις μιας μειοψηφίας μεταξύ των επιστημόνων. Έχει συμβεί μέσα στην ΕΦΣΑ μέσα στη λειτουργία των πάνελ, κάποιες φορές να μην προκύπτει μια γενική συνένεση, μια γενική συμφωνία <clears throat> μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. Και υπήρξαν περιπτώσεις που εκφράστηκαν απόψεις μειοψηφίες από ένα, δύο ή και περισσότερους επιστήμονες στο πάνελ. Παραδείγματος έγινε αυτό για την ευζοία των ζώων και την υγεία των ζώων και επίσης σε μια κοινή γνωμοδότησή μας για την αντιμικροβιακή αντίσταση που μπορεί να μεταφερθεί από μεταλλαγμένους οργανισμούς στο περιβάλλον και επίσης το πάνελ για την υγεία των φυτών. Επομένως, μια τέτοια διαδικασία με απόψεις μειοψηφία είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, δεν είναι αυτόματη η ομοφωνία μεταξύ των μελών του πάνελ. Αν υπάρχουν μειοψηφούσες απόψεις, αναφέρονται πάντα στη γνωμοδότησή μας και φυσικά όλα αυτά είναι ανοιχτά και διαθέσιμα προς το κοινό. Δεν αποκρύπτουμε λοιπόν τέτοιες μειοψηφούσες απόψεις και αυτό είναι γενική γραμμή πλεύσης στο έργο μας. Επίσης, μέσα στα πλαίσια των εργασιών μας, εξασφαλίζουμε το ότι θα πρέπει οι αβεβαιότητες να διατυπώνονται με κάποια σαφήνεια. Δηλαδή, η επιστήμη αφορά και τη δυνατότητα να αμφιβάλλει κανείς και να θέτει ερωτήματα και σε όλους τους τομείς που αναπτύσσουμε την αξιολόγηση των κινδύνων δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι είμαστε βέβαιοι για κάτι. Πολλές φορές δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, πολλές φορές υπάρχουν αμφιβολίες και αβεβαιότητες και εμείς φροντίζουμε πάντα να εκφράζουμε αυτές τις αβεβαιότητες και τις ελλείψεις γνώσης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ε, έχουμε εργαστεί ώστε τα πάνελ μας να έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να εκφράζουν τις αμφιβολίες αυτές. Φυσικά σε ορισμένου τομεί αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Όπως παραγωγή χάρη όταν μιλάμε για νέες τεχνολογίες, όπου μπορεί να είναι μεγάλες οι αβεβαιότητες. Παραγωγή χάρη, όταν είχαμε δώσει μια γνωμοδότηση για την κλωνοποίηση, είχαμε αναφέρει ότι είναι ελάχιστα τα στοιχεία και ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει κανεί σε μια αξιολόγηση κινδύνου παρά το γεγονός ότι είπαμε ότι επί τη βάση των δεδομένων τα οποία ήταν διαθέσιμα και έχοντα εξασφαλίσει ότι εκφράζουμε το υψηλό επίπεδο αβεβαιοτήτων που παραμένουν, είχαμε πει ότι για τα θέματα της ασφάλειας τροφίμων η τεχνολογία κλωνοποίηση δεν ήταν πιθανό να οδηγεί σε προβλήματα. Αλλά είπαμε από την άλλη πλευρά ότι μπορεί η κλωνοποίηση να έχει σημαντικά προβλήματα για την ευζοία των ζώων και την υγεία τους. Εμείς θέλουμε να αμφισβητούμεθα. Η επιστήμη έχει σαν βάση την συζήτηση, το διάλογο και πρέπει κανείς να καταθέτει τις απόψεις του φροντίζοντας την ποιότητα του διαλόγου. Το 863 ε, ε, έγινε ολόκληρη συζήτηση, υπήρξε μια δημοσίευση σχετικά με τη χρήση στατιστικών μεθόδων για την αξιολόγηση κινδύνου των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Μόλις δημοσιεύθηκε η μελέτη αυτή αποφασίσαμε να ξανακάνουμε την έρευνα. Εργαστήκαμε εσωτερικά με τους εμπειρογνώμονες, τους εσωτερικούς αλλά και με εξωτερικούς επίσης στατιστικολόγους έτσι ώστε να δώσουμε στο πάνελ γενετικά τροποποιημένων οργανισμών μια πραγματική αξιολόγηση αυτών των μελετών. Κάναμε συγκρίσεις των δύο στατιστικών μεθόδων αυτή που χρησιμοποίησε η υπηρεσία μας και αυτή που χρησιμοποιήθηκε στο άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε ε, στο ε, γνωστό αυτό επιστημονικό περιοδικό. Και ναι μεν αναγνωρίσαμε ότι η μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό ήταν πράγματι έγκυρη και ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί μεθοδολογικά σαν σωστή. Υπογραμμίσαμε όμως ότι δεν επηρέασε την έκβαση της δικής μας αξιολόγησης, γιατί δεν υπήρξε καμία βιολογική διαφοροποίηση των δύο στατιστικών μεθόδων. Συγγνώμη που μπαίνω σε κάποιες λεπτομέρειες, λίγο τεχνικές, αλλά πρέπει να πούμε ότι εμείς στην υπηρεσία μας δεν φοβούμεθα να αμφισβητηθούμε και να εξετάζουμε νέες επιστημονικές πληροφορίες. Και δεν διστάζουμε να πούμε ότι για κάποια προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται επί μακρόν στην Ευρώπη, ότι μπορεί να υπάρξουν νέοι κίνδυνοι ή να υπάρξουν κάποιες νέες επιστημονικές πληροφορίες που μας οδηγούν στο να αναθεωρήσουμε το καθεστώς ε, των ε, συγκεκριμένων προϊόντων και αυτό έχει τα αρώματα στα τρόφιμα. Συμφωνώ επίσης και όσα είπατε για το περιβάλλον και την αξιολόγηση των κινδύνων για το περιβάλλον. Αυτό δεν είναι άμεση αρμοδιότητα της ΕΦΣΑ. Αλλά παρόλα αυτά είναι ευθύνη μας ε, να ε, υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει η προσπάθεια αυτή. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση. Particularly highlighted the importance of taking care um, Σαν παράδειγμα φέρνω το LN όριζα 62 το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο αξιολογήθηκε σε σχέση με τις περιβαλλοντικές ε, ε, επιβαρύνσεις τις οποίες μπορεί να προκαλέσει. Είπατε ότι δεν είμαστε συστηματικά ενήμεροι και επίσης ε, δεν ολοκληρώνουμε πάρα πολύ συχνά τις μελέτες μας τις 90 μέρες όπου αυτό απαιτείται. Έχουμε προσαρμόσει την μεθοδολογία μας ε, σε σχέση με τη συγκεκριμένη αυτή μέθοδο των 90 ημερών και έχουμε πει εκεί όπου είναι ο, τις περιπτώσεις τις οποίες είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μελέτη μέγιστης διάρκειας 90 ημερών. Δεν θέλω να σας δώσω τώρα περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούμε, αλλά δεν συστήνουμε συστηματικά τις 90 ημέρες για τα γενετικά τροποποιημένα. Και αυτό το κάνουμε υπό το φως ακριβώς των διεθνών ε, επιστημονικών ε, κατευθύνσεων. Μία από τις σημαντικές μας συστάσεις και αυτό δεν το κάνουμε για να ξεφύγουμε από το θέμα της αξιολόγησης κινδύνων. Αλλά υπάρχει το θέμα των ανθεκτικών σε επίπεδο ζυζανιοκτώνων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Απαιτείται να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει μια αυξανόμενη αντίσταση στις ουσίες αυτές από το περιβάλλον. Αν θέλετε να επανέλθω στις ερωτήσεις τις οποίες πιθανώς δεν έδωσα απαντήσεις στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή, αυτός ήταν ο γύρος ε, ερωτήσεων και απαντήσεων. Νομίζω ότι έχετε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Βρισκόσαστε υπό τους προβολείς της δημοσιότητας. Είναι 450 μέλη του προσωπικού σας που είναι υπερήφανοι και χαρούμενοι, αυτό μπορώ να το καταλάβω, διότι το έργο σας για την ασφάλεια των τροφίμων είναι κάτι το οποίο εγώ θεωρώ οπωσδήποτε ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα και να μπορούν οι πολίτες, οι καταναλωτές να νιώθουν ασφάλεια σε σχέση με τα τρόφιμα ότι δεν έχουν επομένω τοξικά προϊόντα, αλλά είναι πάρα πολύ υγιεινά τα τρόφιμα του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε απαντήσει λοιπόν εκτενώ σε όλα τα ερωτήματα. Εμεί ω ε, Προεδρείο, ω ε, συντονιστέ τη Επιτροπή, θα αποφασίσουμε ποιο θα είναι και το άτομο που θα είναι ο σύνδεσμο με τον φορέα σα και θα συνεχίσουμε μάλλον το έργο αυτό τη ε, συνεργασία σα. Μας έχετε προσκαλέσει στην Πάρμα κάθε δύο χρόνια. Πηγαίνουμε εκεί με μια μικρή αντιπροσωπεία. Το 2010 πάλι θα έρθει μια αντιπροσωπεία επιτοπίως για να συναντηθεί μαζί σας. Εγώ σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στο έργο σας και θα ξαναειδωθούμε είτε εδώ στην Επιτροπή μας είτε σε εσάς στο φορέα σας στην Πάρμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μάλλον σύντομη η συνεδρία σήμερα. Εάν δεν διαφωνείτε να προτάξουμε το σημείο 5, γιατί έχω και άλλο ραντεβού και κανονικά έπρεπε να είχα ήδη φύγει. Αλλά δεν πειράζει, ε, παραμένω και με χαρά. Ε, προς, ε, κοίτα για την επιτροπολογία. Το Κοινοβούλιο σε ψήφισμα του κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει την κείμενη νομοθεσία ε, για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να ασκήσει τα δικαιώματά του ε, ε, σύμφωνα με την επιτροπολογία. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Omnibus. Πέντε συγκεκριμένοι, γιατί έχουμε ένα πηγενέλα πολλών εγγράφων και έχουμε μια οδηγία που ασχολείται με την η υγεία των ζώων στο ενδοκινοτικό εμπόριο και μια άλλη οδηγία για την καταγραφή βοηδών και τη σήμανση του βοήου κρέατος. Η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή εδώ είναι η νομική. Εμείς νομοδοτούμε απλώς. Και η γραμματεία και εγώ βρήκαμε όλα αυτά τα σημεία, εννέα τον αριθμό, Και βάζουμε πάντα μια παράγραφο εκεί, ένα εδάφιο, ότι θα πρέπει να ε, χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη διαδικασία κανονισμού, κανονιστική διαδικασία με ε, συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Με έλεγχο δηλαδή. Ε, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να σχολιάσει κανείς εδώ. Εννέα περιπτώσεις σας είπα εντοπίσαμε. Αύριο αποφασίζει η νομική επιτροπή, γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να ψηφίσουμε εμείς σήμερα, για να φτάσει εγκαίρω στη νομική. Ρωτώ, τυπικά, τα μέλη της Επιτροπής έχουν να προσθέσουν ε, και άλλες παραγράφους που ανακάλυψαν στις οδηγίες αυτές. Όχι. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε όλες τις περιπτώσεις μαζί, αν μπλοκ όπως λέμε εδώ, γιατί είναι πάντα το ίδιο αντικείμενο. Όχι! Ξεχωριστά! Καλά τότε. Ε, το υποστούμε και αυτό. Λοιπόν, η τροπολογία αριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Α, βλέπω ότι έχουμε και αντιστάσεις εκεί πίσω. Η τροπολογία υπαριθμών 2. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 3, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το ίδιο για την 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 9. Η 8 συγγνώμη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία για την έκθεση αυτή. Υπέρ. Να μετρήσουμε. Κατά. Απόχες. 26 υπέρ και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία στο θέμα αυτό και Παραδίδω την Προεδρία στην κυρία Κόρνη Λεπάζ για το σημείο υπαριθμών 4 που είναι και το τελευταίο στην ημερήσια διάταξη για σήμερα το απόγευμα. Euh, Καλώς λοιπόν. Έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης για την απόφαση του Συμβουλίου που αφορά την, εκ, την έκθεση των παρατηρημάτων 2 και 3 που αφορούν την αποθήκευση ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακου σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Σύμβαση ως ΠΑΡ. Η εισηγήτρια είναι η Άννα Ροσμπαχ για το έγγραφο αυτό. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Ρόσμπαχ, εφόσον ευαρισκείται να λάβει το λόγο και να μας παρουσιάσει την εκθεσή της. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής μας γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει ΟΣΠΑΡ για τους ε, νέους βουλευτές. Θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για μια σύμβαση για την προστασία του Βόρειου Ατλαντικού, του περιβάλλοντος του Βόρειου Ατλαντικού, όπου συμμετέχουν φυσικά και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1972 δημιουργήθηκε ο φορέας αυτός στο, στο Όσλο, στην Νορβηγία και προστατεύει τους ωκεανούς από την απόρριψη διαφόρων ουσιών και επίσης λαμβάνει υπόψη και τη λειτουργία των υπεράκτιων ε, δραστηριοτήτων. Έχουν συγχωνευτεί οι δύο λοιπόν συμβάσεις που αφορούσαν τα δύο αυτά τμήματα και έχει επίσης διευρυνθεί η σύμβαση αυτή για τα θέματα της βιοποικιλότητας, δηλαδή για δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την ε, ρήπανση και μόνο. Η Φιλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ενωμένο Βασίλειο, κάτω χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία συμμετέχουν στη σύμβαση αυτή για την προστασία του Βορειοατλαντικού, ΟΣΠΑΡ. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, ε, συμμετοχή της Ελβετίας λόγω του Ρήνου, ο οποίος περνάει από την Ελβετία και της Φιλανδίας γιατί μπορούν να περάσουν ρηπαντικές ουσίες στη Βόρεια Θάλασσα. Έχουν συμπεριληφθεί λοιπόν στην σύμβαση αυτή τα παρατήματα 2 και 3 σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ε, ρευμάτων διοξιδίου του άνθρακος στον πυθμένα της θάλασσας. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία στους χώρους οι οποίοι καλύπτονται από τη σύμβαση ΟΣΠΑΡ. Μπορείτε να διαβάσετε τις τροπολογίες λοιπόν στη... οι οποίες θα πρέπει να τύχουν απόφασης. Όσο περισσότερο διαβάζω για το θέμα αυτό, τόσο περισσότερα ερωτήματα θέτω στον εαυτό μου και όσο περισσότερο βλέπω το χάρτη των περιοχών για τις οποίες αναφερόμαστε, τόσο πιο σαφές γίνεται σε μένα ότι ο τομέας, ότι ο χώρος του κεντρικού Ατλαντικού περιλαμβάνεται στο, στην απόφαση αυτή. Και εδώ τίθενται θέματα συνείδησης για τους πολιτικούς. Υπάρχουν συγκεκριμένε μελέτες σε αυτή την περίπτωση. Προσπάθησαν και σεισμολόγοι να ελέγξουν την ασφάλεια της εναπόθεσης αυτών των αποβλήτων και τίθενται πάρα πολλά προβλήματα για τα πυρηνικά αποβλήτα τα οποία δεν έχουν τύχει απάντησης μέχρι τώρα. γιατί ξέρετε ότι αν τυχόν ε, υπάρξει η σπίδηση ύδατος σαν παράδειγμα, ε, τότε μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον πολύ σοβαρά προβλήματα. Και αν υπάρξουν κατακριμνήσεις βυθού, θα δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα και πιθανότητα ατυχημάτων θα είναι υψηλή και ποιος θα είναι υπεύθυνο ε, για τα ατυχήματα αυτά, ποιος θα είναι σε θέση να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανώς τέτοιων καταστροφών. Ιδιαίτερα αν συμβεί κάτι σε διεθνή ύδατα. Τι θα περιμένουμε, θα περιμένουμε να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο σενάριο στο οποίο θα έχουμε καταλήξει ή μήπως θα περιμένουμε να συμβεί κάτι πρώτα για να αντιδράσουμε εκ των υστέρων. Άκουσα ότι η διαδικασία αποθήκευσης είναι κάτι το οποίο κοστίζει μάλιστα πάρα πολύ. Ε, ε, ε. Συνεπώς τι γίνεται και με τους, την ασφάλεια των εργαζομένων που ασχολούνται με την εναπόθεση των αποβλήτων. Είναι κάτι το οποίο καλύπτεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κάποιε διεθνείς συμβάσει. Όλες αυτές οι απορίες είναι συμπτωματικές θα έλεγα τη κατάστασης ε, με την οποία, σύμφωνα με την οποία λειτουργεί η κοινωνία μας σήμερα. Το μοναδικό πράγμα στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας να αντιπροσωπεύσει ένα παράδειγμα για άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και η Ρωσία. Αλλά δυστυχώς φοβούμεθα ότι όπως και εμείς και οι χώρες αυτές δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να δημιουργήσουμε τα συστηματικά μέτρα ελέγχου τα οποία απαιτούνται για να τελειώνουμε. Η λύση η οποία προτείνεται είναι η καλύτερη και για το διοξίδιο του άνθρακα ή μήπως θα πρέπει ε, καλύτερα να στρέψουμε τους ερευνητές να αναζητήσουν διαφορετικές λύσεις για την αποθήκευση ε, του διοξιδίου του άνθρακα, διότι το θέμα είναι ότι η αναζήτηση θα πρέπει να στραφεί περισσότερο στην εκ νέου χρήση του διοξιδίου αυτού. Σας ευχαριστώ κύριε Ρόσμπαχ. Σας ευχαριστώ που απευθύνατε έκκληση στις γνώσεις μας αλλά και στη συνείδησή μας. Γιατί πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και αναλαμβάνουμε ευθύνε σε σχέση με τα πράγματα για τα οποία είμαστε πράγματι μακριά από να γνωρίζουμε τις συνέπειες τους. Και σας ευχαριστώ που μας το θυμήσατε αυτό. Θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Μορκουνάιτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα να παρουσιάσω ποια είναι η δική μας θέση για το έγγραφο αυτό στη σημερινή συζήτηση. Το ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέση σαν στόχο του σε σχέση με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή το να μειωθεί η αύξηση της θερμοκρασίας και να παραμείνει μέσα στα όρια των δύο βαθμών. Θέλουμε επίση να μειώσουμε τα αέρια θερμοκηπίου κατά 30%. Η αποθήκευση του διοξίδιου του άνθρακο σε φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς που προβλέπεται στα παρατήματα 2 και 3 της Σύμβασης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος είναι ένα βήμα προς τα εμπρός σε τεχνολογική, από τεχνολογική άποψη για να απαλύνει τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Μετά από την υπογραφή αυτής της σύμβασης έχει γίνει δυνατό, χάρη στην βελτίωση τεχνολογίας, να υπάρχει συγκράτηση του διοξιδίου του άνθρακος και αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς στον πυθμένα της θάλασσας. Επομένως, απομονώντας το διοξίδιο του άνθρακος αυτό από το γενικό κύκλωμα κυκλοφορίας στην γη και στην ατμόσφαιρα. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει αυτές τις αλλαγές, τα παρατήματα, τονίζοντας πάντα ότι η σύμβαση, σύμβαση βασίζεται στην ιδέα ότι πριν ληφθεί μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες να υπάρξει ρήπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον και αντικές συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αποτρέψουμε τέτοιες αντικές συνέπειες. Εγώ έρχομαι από τη Λιθουανία, μια χώρα που βρίσκεται στη Βαλτική, που είναι ίσως η πιο ρηπασμένη θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χώρα μου, όπως και οι όμορες χώρες, γνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για το περιβάλλον λόγω των ε, τοξικών υλικών που βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας. Όταν λοιπόν υπάρχει πρόταση να δημιουργηθεί ο αγωγός North Stream, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή κατασκευής μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές οικολογικές καταστροφές, θέλω να χαιρετήσω τις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος, και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές, αλλά μόλον τούτο θέλω να υπογραμμίσω την μεγάλη ευθύνη που θα πρέπει όλοι να επομιστούμε για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα πρέπει να δράσουμε με ένα πάρα πολύ προσεκτικό και επάγρυπνο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και την προστασία του περιβάλλοντο. Κύριε Σασένης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κάθε χρόνο αναγνωρίζουμε και περισσότερο τη σημασία των φυσικών οικοσυστημάτων και της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Και έχουμε και προτάσεις για τεχνικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Στοιχώς, βλέπουμε πάντα ότι οι τεχνικές λύσεις έχουν και παρενέργειες προς το περιβάλλον, αρνητικές παρενέργειες. Μιλάμε τώρα για την συγκράτηση και την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακος. Μιας τεχνολογίας η οποία δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα σε πραγματικές συνθήκες. Μπορεί να έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα, αρνητικά για το περιβάλλον και για τους ωκεανούς. Γι' αυτό το λόγο Αντίστοιχα σχέδια δοκιμάστηκαν στη Γερμανία και στην Ολλανδία, αλλά εκεί οι οργανώσεις των πολιτών αντιτάχθηκαν γιατί θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον από απρόβλεπτα αποτελέσματα. Θέλουμε τώρα να δοκιμάσουμε κάτι στον Ατλαντικό, εκεί που δεν υπάρχει η κοινωνία των πολιτών η οποία να αναχαιτήσει αυτά τα σχέδια. Επομένως, εμείς θα πρέπει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσουμε πώς θα αποτρέψουμε αρνητικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε και τα αποτελέσματα αυτού του σχεδίου για τη βιοπικιλότητα, αλλά και το σωρευτικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την προστασία του Ατλαντικού. Και θα πρέπει να βρούμε <clears throat> τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις ε, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και συγχρόνως να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση της ευκαιρίας που μας δίνει στη της Κοπενχάγης, γιατί μας έχουν επικρίνει, γιατί δεν έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να προσαρμοστούμε σε μια χωρίς άνθρακα οικονομία στον πλανήτη μας. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν τα καλύτερα κίνητρα για να μειωθεί και η παραγωγή αλλά και η κατανάλωση ενέργειας και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το σχέδιο αυτό δεν δίνει ένα λανθασμένο μήνυμα που αντίκειται προς τα κίνητρα τα οποία θέλουμε να παρέχουμε εμείς και ότι δεν θα παίξει το ρόλο αντικινήτρου για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρωπου. Ευχαριστώ, Chris Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήμουν εισηγητής που συνόδευσε αυτή την οδηγία στο Κοινοβούλιο πέρυσι. Και μερικά από τα επιχειρήματα που ακούσαμε τώρα είναι επανάληψη των περσινών συζητήσεων. Ποια είναι η προτεραιότητα παραμένει ίδια για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. 25% όλων των εκπομπών ε, στην Ευρώπη προέρχονται από τον άνθρακα. Και μετά έχουμε τα ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο και ε, φυσικό αέριο που παράγουν ηλεκτρισμό. Και το 40% όλων των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μπορούν να μετριαστούν με τη τεχνολογία αυτή. Στην τελευταία συνεδρίαση ακούσαμε ότι η Κίνα επεκτείνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτές οχριούν μπροστά στα νέα ε, θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Φτιάχνουν ένα εργοστάσιο κάθε λίγες μέρες. Και διεθνείς οργανισμοί, ε, υπολογίζουν ότι τα επόμενα 20 χρόνια θα αυξηθεί η κατανάλωση άνθρακα κατά 60%. Όσο και αν επενδύουμε σε ανανεώσιμες πηγές ή και σε πυρηνική ενέργεια, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τον άνθρακα και τα ορυκτά καύσιμα. Χωρίς, αν ε, δεν χρησιμοποιήσουμε την ε, δέσμευση και αποθήκευση ε, διοξιδίου του άνθρακα είναι αποσπασματικέ οι προσπάθειες. Δεν έχει γίνει ποτέ προσπάθεια συγκέντρωσης για ε, να ε, γίνει κάποια κοινή προσπάθεια σε εργοστάσια μεγάλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει συστάσεις ε, γύρω στα έξι προγράμματα, ερευνητικές προσπάθειες θα ενταχθούν και στο σχέδιο της ανάκαμψης. Μέχρι 180 εκατομμύρια ευρώ, λέει το πρακτορείο Reuters, ότι θα φτάσουν οι ενισχύσεις ε, Πολωνία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, κάτω χώρες και Αγγλία. Και τέλη Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, ελπίζουμε, θα συμφωνήσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν τις επόμενες επενδύσεις που απελευθέρωσε το Κοινοβούλιο της Πιστώσης πέρυσι ε, και αναφέρομαι στα δικαιώματα εκπομπών και στα έσοδα από την εμπορία. Μέχρι 6 δισεκατομμύρια μπορούμε να φτάσουμε στη χρηματοδότηση για ε, προγράμματα επίδειξη τεχνολογία. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω το πακέτο αυτό να συμφωνηθεί τέλη Οκτωβρίου και να μπορέσουν να προχωρήσουν τα ερευνητικά σχήματα αυτά. Η συγγήτρια ανέφερε κάποια θέματα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια οδηγία δηλαδή που λέει ότι όταν υπάρχει άδεια για την ε, αποθήκευση δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διαρροή, ούτε καν υπόνη, υποψία διαρροής για να ε, δοθεί έγκριση. Και επίσης να έχουμε και ε, ε, κάποια πρόνοια για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και φερεγγιότητα. Εδώ μιλάμε για το βορειοανατολικό Ατλαντικό. Το ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πολύ μακριά από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται εδώ με την ευθύνη. Ε, δεν έχω καταλάβει προς τα που πηγαίνουμε για να βεβαιωθούμε ότι η νομοθεσία μας εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο και εκεί στα βάθη του ωκεανού και τόσο μακριά. Και τέλος, ε, συμπερασματικά θέλω να πω ότι η πρόταση αυτή φιλοδοξεί να εξασφαλίσει μια αρμονία ε, μεταξύ των δικών μας κανόνων και εκείνων του ΟΣΠΑΡ. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε τα, ε, τις ίδιες ρυθμίσεις και διατάξεις για την ασφάλεια και εμείς και η Σύμβαση ΟΣΠΑΡ. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να ξεφύγει από το δοκιμαστικό στάδιο αυτή η τεχνολογία και να ε, μπει στο στάδιο της επίδειξης, να αναπτυχθεί πλήρως. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ακούστηκε επίσης ότι είναι σαν να θάβεις απόβλητα. Ναι, εντάξει. Το διοξείδιο του άνθρακα ε, απαντά και στη φύση. Όταν κάνεις ε, ε έρευνες για πετρέλαιο, καμιά φορά πέφτεις και σε διοξείδιο του άνθρακα. Και βέβαια δεν είναι μακροπρόθεσμη λύση για το πρόβλημά μας αυτό, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο το συντομότερο, το συντομότατο να αναπτύξουμε αυτές τις τεχνολογίες για να καταπολεμήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Άμα τα θάψουμε εκεί στα βάθη του ωκεανού, ε, τόσο βαθιά, ε, σε κάποια, ε, σε κάποια φάση θα στερεοποιηθεί αυτό και θα μείνει στο φλοιό της γης. Και δεν θα είναι στην ατμόσφαιρα να επιβαρύνει και να απειλεί τις επερχόμενες γενναίες. Euh, Ευχαριστώ, Chris Davis. Η κυρία Ντεμπρούν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλη κατανόηση και συμπάθεια βλέπω τις ερωτήσεις πολλών συναδέλφων που μίλησαν προηγουμένως και πολλές θα τις είχα κάνει και εγώ και έτσι με μεγάλο σθένος όταν ήμουν σκιώδης εισηγήτρια για το τμήμα της οδηγίας που μας απασχολεί σήμερα εδώ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμο να κοιτάξουμε αυτό που είπε ο Chris Davis. Και αναφέρουμε κυρίως αυτό που είπε στο τέλος. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Έχουμε και οδηγία. Ε, τώρα τι συζητάμε. Είναι η δυνατότητα που έχουμε ε, να κάνουμε την οδηγία που ήδη ψηφίσαμε νομοθεσία, να τη βάλουμε σε μία σύμβαση. Αυτό λέει. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι όμως για να ξέρουμε ότι αυτό που ψηφίσαμε πέρσι με όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις και δικλίδες, με όλη αυτή τη φασαρία που έγινε και τη μάχη για να καλύψουμε ε, κάπου τα στοιχεία ασφαλής, να μην τα χάσουμε κάπου στον δρόμο ε, μένοντας στη σύμβαση Ωσπαρ. Βέβαια, ξεπερνάει την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, αυτή η σύμβαση, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι ήδη στις προδιαγραφές ασφαλείας και οι διατάξεις. this... Να βεβαιωθούμε λοιπόν ότι τώρα είμαστε σε θέση να περάσουμε και διεθνώς αυτό που ψηφίσαμε πέρσι στην οδηγία. Και θα πρέπει απολύτως να ευθυγραμμίζεται με την οδηγία αυτή. Και για την ασφάλεια και για την ευθύνη και για την φερεγγιότητα. Και θέλω κάπως αυτό να μας το διευκρινίσετε. Je Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σνέλχαρτ έλαβε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στην προηγούμενη θητεία Είχαμε συζητήσει ιδιαίτερα για την τεχνολογία συγκράτησης και αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακος και όπως είπε και ο Κριστέβη. καταλήξαμε σε μια απόφαση η οποία ήταν, πιστεύω, τελής. Νομίζω ότι υπήρχαμε, υπήρχε στην αρχή ένα μεγάλο μέρος αμφιβολιών για την τεχνολογία αυτή, για τη συγκράτηση και την αποθήκευση του διοξείδιου του άνθρακος. Έδειξαν όμως οι συζητήσει ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε τον αγώνα για την κατά της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την τεχνική, θα πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε το διοξείδιο του άνθρακος δεν εκφεύγει στην ατμόσφαιρα. Όταν λοιπόν θέλουμε κάτι τέτοιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα αυτή να χρησιμοποιήσουμε ως φορέα παραγωγής ενέργειας τον άνθρακα μαζί με τις ανανεώσιμες ενέργειες. Αυτό όμως προ... προϋποθέτει ότι θα έχουμε τρόπους να μπορούμε να αποθηκεύουμε ασφαλώς το διοξείδιο του άνθρακος και να το βγάζουμε από την κυκλοφορία. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός ε, δρόμος που ακολουθούμε. Η χώρα μου, η Γερμανία, προβλέπει να κάνει ένα σχέδιο επίδειξης μέσα στο οποίο θα εφαρμοστεί πράγματι αυτή η τεχνολογία και πράγματι βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο της επίδειξης βέβαια. Τίθεται προφανώς το θέμα του κόστους. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να ε, καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή η τεχνολογία έχει προχωρήσει σημαντικά. Επομένως, όταν υπάρχει η καύση άνθρακος, αυτό δεν οδηγεί αδύρυτα σε εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος. Μπορούμε λοιπόν για να χρησιμοποιήσουμε τον άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας είναι απαραίτητο να βρούμε τους τρόπους να αποθηκεύουμε το διοξίδιο του άνθρακος και θα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και στην περίπτωση εδώ της ΟΣΠΑΡ ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογικές βελτιώσεις για να πετύχουμε το στόχο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αν όμως καθυστερούμε, αν απορρίψουμε αυτή την αλλαγή, χάνουμε αυτή την ευκαιρία. Χάνουμε μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε το θέμα του διοξιδίου του άνθρακος. Εγώ νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να δεχτούμε αυτή την αίτηση που είναι ενώπιόν μας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόντι. Ήδη είχαμε τη δυνατότητα στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο να συζητήσουμε σε βάθος τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι η σωστή λύση. Γιατί το 1 τρίτο της ενέργειας που παράγεται θα πρέπει να στοχεύει στον διαχωρισμό, στη συμπίεση και στην αποθήκευση του διοξιδίου. Συνεπώς αντικειμενικά θα έλεγα, η ιδέα αυτή Ενό είδους χωματερή στη θάλασσα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απορρίψουμε ουσιαστικά γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί. Ε, πάντως φαίνεται ότι θα προχωρήσει η ιστορία αυτή. Δεν συμφωνώ πάντως και με την χρηματοδότηση που θα πρέπει να δώσουμε. Νομίζω ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να προέλθει κυρίως από το σύστημα εμπορίας ρήπων. Γιατί μακροπρόθεσμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να επιδιωχτούν. Πέραν του γεγονότος της ύπαρξης μιας μορφής θα έλεγα συγκέντρωσης ουσιαστικά του διοξιδίου του άνθρακα που δεν στοιχειοθετεί εναπόθεση του άνθρακα αλλά φυτικής προέλευσης άνθρακας ο οποίος θα μπορούσε να αναμειχθεί με το χώμα και αυτό να βελτιώσει και την οικονομική εκμετάλλευση των υδάτων και να καταστήσει πιο γόνιμα τα συγκεκριμένα εδάφη. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια δραστήρια και ενεργή παρακράτηση του διοξιδίου του άνθρακα με μια δεύτερη χρήση. Και αυτό θα πρέπει να επιδιώξουμε, αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε. Πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία αφορά στην ανάκτηση του διοξιδίου του άνθρακα και στην εκ νέου χρήση του για θετικούς λόγους και όχι να ακολουθήσουμε την απλή εναπόθεση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόντι. Δεν υπάρχουν ε, άλλοι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο και θα δώσω εκ νέου το λόγο. Α, όχι, πρέπει να δώσω το λόγο και στην Κομισιόν, αν το θέλει. Κύριος Κάρλος Δεχοσέ Γκαρσία. Thank you. Ευχαριστώ. Η Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μερικές απαντήσεις μόνο. Η δέσμευση και αποθήκευση ε, του διοξιδίου του άνθρακα είχε προταθεί ως ε, τεχνολογία συγκράτησης ε, της υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής, αλλά το θέμα είναι αν έχουμε νέα στοιχεία, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκρινε το 2009 ε, τον Ιούνιο την Οδηγία 31 και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν νέα <laughs> στοιχεία. Είναι ένα σαφές νομικό πλαίσιο που χρειάζεται για να ε, καλύπτονται και οι κίνδυνοι. Όπως είπε και ο Κρίς Ντέιβις. θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει ε, σοβαρός κίνδυνος διαρροής. Εάν καμιά φορά ε, παρόλες τις ε, επιφυλάξεις και ε, παρελπίδα έχουμε διαρροή διοξιδίου του άνθρακα, καλύπτεται από άλλη οδηγία. Επίσης έγινε λόγος για την περιβαλλοντική ευθύνη και το καθεστώς αυτό το οποίο ήδη ισχύει και επιπλέον υπάρχει και το σύστημα εμπορίας εκπομπής ρήπων και σε περίπτωση ακριβώ διαρροών πρόκειται για το υδάτινο περιβάλλον για την ατμόσφαιρα. Τα κράτη-μέλη ε, γνωρίζουν την νομοθεσία αυτή, την εφαρμόζουν και τα περισσότερα συμβαλόμενα μέρη της ΟΣΠΑΡ είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υπόλοιπα που βρέχονται από ε, τον Ατλαντικό είναι ε, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και θα συμπεριληφθεί η οδηγία αυτή για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα ε, στις συμφωνίες που έχουμε. Ε, το θέμα είναι λοιπόν κατά πόσο αυτά που ενέκρινε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το καλοκαίρι μπορούν να μεταφερθούν εκεί. Βεβαίω, εμείς απαντάμε καταφατικά, θα πρέπει να παραμείνει όπως έχει η απόφαση του Ιουνίου. Να σας ε, διευκρινίσω λίγο το πεδίο εφαρμογής που ρώτησε ο Κρις Ντέιβις, η οδηγία αφορά τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών ή τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες που είναι 200 ναυτικά ε, μίλια για τα παράκτια κράτη-μέλη, αλλά και την υφαλοκρηπίδα των κρατών μελών. Άρα, καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Βόρειας Θάλασσας, όπου ε, μπορεί ε, να υπάρξει τέτοια οικονομική δραστηριότητα για το διοξίδιο του άνθρακα. Το θέμα ε, της δοκιμασμένης τεχνολογίας και πώς αυτή μεταφέρεται, έχει δίκιο ο Chris Davis. Είναι πολύ λίγα τα παραδείγματα που εφαρμόζονται, αλλά από τα καλύτερα που έχουμε είναι σε γεωλογικό σχηματισμό κάτω από το βυθό της θάλασσας για 10 χρόνια περίπου ένα εκατομμύριο τόνους διοξιδίου του άνθρακα τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν αποθηκευτεί ε, σε ένα βυθό που δεν ε, ε, είχε αυτό καμία παρενέργεια, είτε πρόκειται για το φυσικό περιβάλλον, είτε για τον άνθρωπο. Τώρα έχουμε το πρόγραμμα ανάκαμψης που χρηματοδοτεί τις επιδείξεις. Έχουμε και τα δικαιώματα από την εμπορία εκπομπών και γενικότερα πείρα για να επιβεβαιώσουμε το, ότι είναι ασφαλές να αποθηκεύονται έτσι ε, ε, ε, αυτά τα, αυτό το διοξείδιο του άνθρακα. Τώρα, ρωτήσατε τι γίνεται διεθνώς. Και ο Chris και άλλοι είπαν ότι είναι σχεδόν αδιανόητο να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή χωρίς να δούμε τι γίνεται ε, σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, μεγάλες αναπτυσσόμενες αναδυόμενες χώρες με τα ορυκτά καύσιμα. Ε, αυτό το θέμα της δέσμευσης και αποθήκευσης οξυδίου του άνθρακα είναι σημαντικό. Ε, πρέπει να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο και το έχουμε στην Ευρώπη με πολύ καλά προηγούμενα, με πολύ καλούς κανόνες για διεθνή εφαρμογή και θα το προτείνουμε και στις διαπραγματεύσεις της Κοπενχάγης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ο κύριο Μπέρο Γκαρσία βλέπω ότι δεν θέλει να παρέμβει. Ξαναδίνω λοιπόν το λόγο οριστικά στην κυρία Ρος Μπαχ. ευχαριστώ όλους για τα θετικά σας σχόλια. Σας ευχαριστώ επίσης για τις γνώσεις τις οποίες μας μεταδώσατε. Παρ' όλα αυτά πρόκειται ε, για κάτι το εντελώς καινοτόμο για μένα βέβαια, αλλά κάποιες περισσότερες πληροφορίες μετά τις παρεμβάσεις σας τις έχουμε. Εξεπλάγιν, βλέποντας ότι το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας μου επηρεάζεται από την υπόθεση αυτή το βόρειο-δυτικό τμήμα, φτάνει μέχρι τη Γρυλανδία ουσιαστικά και είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι μια περιοχή η οποία σίγουρα θα θυγεί από την εφαρμογή του προτινόμενου συστήματος. Νομίζω ότι μια πολύ μεγάλη περιοχή της γης από το Βόρειο Πόλο μέχρι το Γιβλαρτάρ θα επηρεαστούν αρνητικά. Θυμίζω επίσης ότι συμπεριλαμβάνονται περιοχές όπως η Βαλτική θάλασσα με πολύ ειδικά χαρακτηριστικά και όταν υπάρχει ένα πολύ θερμό καλοκαίρι ε, ξέρετε ότι προκαλούνται πολύ έντονες καταστροφές στην οικολογική ισορροπία αυτών των θαλασσών. Και αυτό προστίθεται βέβαια στις ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ισορροπία στις θάλασσες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, ανάγκη να οδηγηθεί σε μια πραγματική λύση διαρκή και αυλαβή για το περιβάλλον για, αυτά τα, για αυτές τις ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό παραμένει σαν αίτημα, αλλά πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι για το τι πράγματι ισχύει στον βυθό των θαλασσών και ειδικά για τη συγκεκριμένη περιοχή, τον βορειοδυτικό Ατλαντικό, α, ίσως να μην είναι η καλύτερη, αλλά από την άλλη σαφώς και υπάρχει ανάγκη να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον με το διοξίδιο του άνθρακα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση ρεαλιστική. Δεν αρκεί ε, με ένα ευχολόγιο, δεν αρκεί ένας κατάλογος επιθυμιών πρέπει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν το περιβάλλον. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Συνάδελφοι, νομίζω ότι είχαμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση γύρω από το κείμενο αυτό. Σας θυμίζω επίσης ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 9η Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα γίνει από τις 3 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου και η τελική ψήφο στην Ολομέλεια μάλλον το Δεκέμβριο. Σας ευχαριστώ. Τέλος των εργασιών για σήμερα.